Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τώρα ε, κοντεύει να τελειώσει η Ολομέλεια, σε ένα-δυο λεπτά και θα τελειώσει, επομένως καλό είναι να ξεκινήσουμε, γιατί ήδη πέρασε η ώρα. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον ε, ε, ε, ο κύριο Μάρου Σεύκοβιτς, Επίτροπο και μελλοντικό αντιπρόεδρο, υποψήφιο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αυτή την τελευταία ακρόαση για φέτος. Εδώ υπάρχουν τα μέλη δύο επιτροπών, Ήτρα και Ένβη και μια και βλέπω ότι είναι πολύ οι παριστάμενοι, ε, καλό θα ήταν να κάνουμε φαίνεται τέτοιε κοινέ συνεδριάσεις και εκτός ακροάσεων. Εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να σας ε, ε, καλωσορίσουμε εδώ. Ε, και να καλωσορίσουμε και τους ε, όσους την παρακολουθούν γιατί είναι μια ανοιχτή ακρόαση. Έχουμε εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, επίσης ε, εκπροσώπους από τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσω διαδικτύου αυτήν την ακρόαση, μέσω του site του Κοινοβουλίου. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους. Κύριε Σεύκοβιτς. Ήδη ε, είχατε μια ακρόαση ε, ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών ε, για την θέση του Επιτρόπου Μεταφορών και Εμπορίου. Οι δύο επιτροπές απεφάνθησαν ότι ο κύριος Σεύκοβιτς ε, έχει όλα τα προσόντα τα οποία χρειάζονται ε, για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στην ε, Κομισιόν. Επομένως, εμείς σήμερα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα νέα ε, χαρτοφυλάκια του ε, Επιτρόπου ε, Σεύκοβιτς όσον αφορά την ενέργεια. Βεβαίως η Επιτροπή μας ασχολείται ιδιαίτερα με την ενέργεια, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια της ενέργειας, την χρήση, την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς επίσης και την ε, προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας. όλα αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα οπωσδήποτε ε, θα αποτελέσουν προτεραιότητες ε, για την επόμενη ε, θητεία και τα μέλη της Επιτροπής μας περιμένουν να δουν τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Εύκοβιτς θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και, τα, και τις προκλήσεις. Έχετε λάβει ένα έγγραφο εκ των προτέρων συγκεκριμένα το mission letter του ε, κυρίου Σεύκοβιτς, υποψηφίου για τα θέματα ε, ενέργειας. Έχετε λάβει το CV του, το βιογραφικό του, έχετε λάβει επίσης το έγγραφο με, τα, ε, με τη δήλωση συμφερόντων του, καθώς επίσης και το ερωτηματολόγιο στο οποίο έχει απαντήσει. Επίσης η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, Γιούρι, Ε, είχε συνεδρίαση σήμερα στις 6 και δεν έχουμε ακόμα λάβει... Α, το λάβαμε. Λάβαμε την επιστολή και από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ναι, τα, τα, πριν από 2-3 λεπτά τη λάβαμε την επιστολή. Και θα την μοιράσουμε την επιστολή αυτή. και αύριο το πρωί θα συζητηθεί στην ε, συνεδρίαση που θα έχουν οι συντονιστές μας, ε, συνεδρίαση αξιολόγησης. Ο συμπρόεδρος Λαδία, παρακαλώ, μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Μπούζεκ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο και ε, υποψήφιο Αντιπρόεδρο για τα θέματα της ενέργειας, ε, τον κύριο Σεύκοβιτς. Ε, γνωρίζουμε την πορεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας, την διπλωματική του πορεία. Το 2004 ήταν ε, μόνιμος αντιπρόσωπος της Σλοβακίας παρά την Ευρωπαϊκή Ενώση επίσης ε, ασχολήθηκε με θέματα ε, αθλητισμού, νεότητας και πολιτισμού στην Κομισιόν μέχρι να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των ε, διαθεσμικών οργάνων στην Επιτροπή Μπαρόζο 2. Το 2014 το Μάιο εξελέγει βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, Περιβάλλοντος και έχω τη μεγάλη αυτή τιμή και βεβαίως είμαστε ιδιαίτερος, δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία πρόκειται ο πρόεδρος Σεφκοβιτς να αναλάβει. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος περίμενε εδώ και πολύ καιρό αποτελεσματική και φιλόδοξη πολιτική περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη οικονομίας, μιας οικονομίας πράσινης και αηφόρου ε, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Ο ε, Επίτροπος ε, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης που θα είναι μακρόθωρη από τη μία και αηφόρος από την άλλη. Επομένως χρειαζόμαστε μια κοινή, ενωμένη και ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν και της διάσκεψης κορυφής των των Παρισίων του 2015 εν ώψη όλων των διακυβευμάτων και των μελλοντικών συμφωνιών όπου θα πρέπει να εκπροσωπεί με ισχυρό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ε, να αναπτυχθεί η πράσινη οικονομία και να γίνει η Ευρώπη η ηγέτιδα όσον αφορά την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως εν ώψη του ορίζοντα 2030 θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω ότι ε, για να μπορέσουμε να ε, κάνουμε ε, μια καλή πράσινη οικονομία και να είναι αηφόρα και βιώσιμη θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε ένα νέο σύστημα ανταλλαγής ρήπων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε, περιμένουμε να ακούσουμε μεγάλη προσοχή αυτά που θα μας πείτε. Ξαναδίνω το λόγο στον συνάδελφο Μπούζεκ. Λοιπόν, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο ε, κύριος Εύκοβιτς θα κάνει μία εισαγωγή 13 λεπτών και μετά 5 λεπτά ε, στο τέλος θα ξαναμιλήσει. Μετά την εισαγωγή του ε, κυρίου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι ήδη και τώρα Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε χρόνο για 41 ερωτήσεις από τους ε, βουλευτές. Η, ομάδα FDD δεν έχει δώσει ερωτήσεις. Τρία λεπτά θα έχει κάθε ερώτηση. Ένα, δύο λεπτά η ερώτηση, ένα η απάντηση ping-pong σύστημα δηλαδή. Και θα έχουμε τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων ε, στην αρχή και τα υπόλοιπα βάσει του, 6, του κανόνα 662. Παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε όλο το χρόνο ομιλίας. Θα έχουμε ανοχή 10 ε, δευτερολέπτων για τον ε, Επίτροπο και 5 για τα μέλη. Μετά από αυτό το όριο ανοχής θα κλείνει το μικρόφωνο δυστυχώς. και πριν από το τέλος του κάθε χρόνου ομιλίας, 10 ε, δευτερόλεπτα, θα αναβοσβήνει ένα φωτάκι. Διερμηνία υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, αλλά παρακαλώ πολύ να θυμάστε ότι δεν πρέπει να μιλάτε γρήγορα, γιατί χρειαζόμαστε ε, καλή διερμηνία αποτελεσματική προς 22 χώρες. Κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε υποψήφιε ε, για τη θέση του Αντιπροέδρου, παρακαλώ πολύ σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές κυρίες και κύριοι, το 2010 ο Γέρζι Μπούζεκ δήλωσε μαζί με τον Ζακ Ντελόρ και παραθέτω χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε την ενέργεια. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή και πιο δυνατή ενεργειακή πολιτική. Στις, ε, στους πολιτικούς προσανατολισμούς του, ο ε, νέος πρόεδρος Jean-Claude ε, βασίστηκε σε, αυτήν, σε αυτό το όραμα έτσι ώστε να αναφέρει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ανεκτική, ανθεκτική όσον αφορά την ενέργεια και να έχει ε, πολιτική ελπιδοφόρα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Ε, στο Lettre de που μου απίφθινε ε, μου Je suis très fier. Επιφόρτησε υπό την ένταση βεβαίω τη δικιά σα σύμφωνη γνώμη να ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Είμαι, είναι τιμή και χαρά ε, για, που μου απέφθηνε αυτή την ε, επιφόρτιση. Οι πολιτικέ ενέργεια και κλιματική αλλαγή ε, βεβαίω βρίσκονται στι πρώτε θέσει τη πολιτική ατζέντα. Σήμερα η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο άμεσε ενεργέ προκλήσει. Πρώτα απ' όλα ε, να ε, διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια, κυρίω στα πλαίσια τη κρίση μεταξύ τη Ρωσία και τη Ουκρανίας, ενώ από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ε, ε, καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ. στην προηγούμενη μακρόαση τόνισα ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από την κατάρρευση του σιδερού παραπετάσματος και 10 χρόνια από την ε, προσχώρηση της χώρας μου και των χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσε τέλος στον τεχνητό αυτό χωρισμό της Ευρώπης. Είναι σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας ενεργειακής υποδομής αυτή είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει μονάχα την οικονομική θεώρηση. Με τα γεγονότα των τελευταίων ετών φαίνεται ότι είναι μια τεράστια προτεραιότητα σε επίπεδο στρατηγική και ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι αυτό το θέμα θα είναι μια πραγματική προτεραιότητα για μένα και θα το αναλάβω με, μεγάλη, με μεγάλο αίσθημα ευθύνη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ε, βουλευτές, και εγώ ήμουνα Υποψήφιο σε ευρωεκλογέ και εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να μπορούν οι πολίτες να έχουν θέσει εργασίες, να μπορούν να έχουν οικονομική ανάπτυξη και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πλήρως την πιο δύσκολη κρίση που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τους πολίτες μας είναι το θέμα των ενεργειακών τιμών. Ο χειμώνα του 2009 είναι ένα χειμώνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ γιατί η Σλοβακία ουσιαστικά βυθίστηκε στο σκοτάδι. Για πάνω από δύο εβδομάδε δεν λειτουργούσε η οικονομία. Μόνο τα νοσοκομεία και τα νοικοκυριά είχαν ενέργεια ενώ είχαν κλείσει τα εργοστάσια. Ξέρετε βέβαια ότι δεν ήταν μοναδική χώρα η Σλοβακία σε αυτή την κατάσταση χωρί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την άμεση ευρωπαϊκή αρρωγή. Οι συνέπειε αυτών των γεγονότων θα μπορούσαν να είναι πραγματικά φρικτές. Γι' αυτό είναι το πραγματικό μας καθήκον, το επιτακτικό μας καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας θα αντιμετωπίσουν και πάλι τέτοιες καταστάσεις. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε αντλήσει διδάγματα από αυτή την κρίση. Όπως έδειξαν οι δοκιμασίε αντοχής για το φυσικό αέριο, είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την Ουκρανία με ανάδρομη ροή φυσικού αερίου από τη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Και αυτό είναι πολύ σωστό γιατί βλέπουμε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την παροχή φυσικού αερίου σαν όπλο άσκηση πίεση και ω πολιτικό όπλο εναντίον τη Ουκρανία και άλλων χωρών που θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Αυτό είναι απόλυτα παράδεκτο. Εάν αποκομίσω την υποστήριξή σα, θα αντιμετωπίσω το θέμα τη ενεργειακή ασφάλεια και θα του δώσω την πρωταρχική προσοχή μου, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. <clears throat> Οι δοκιμασίες αντοχής έδειξαν ότι μπορεί να περιοριστεί ο αντίκτυπος μιας μείωσης της ροής ε, φυσικού αερίου αν εργαστούμε όλοι από κοινού και δεν έχουμε καθαρά εθνικές προσεγγίσεις. Έχει έρθει η χρονική στιγμή για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Για αυτού οι οποίοι είχαν σκεπτικισμό για τα θέματα αυτά, θα του θυμίσω ότι πριν από 70 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απλώ ένα όνειρο. Ήταν αδιανόητο πριν από 25 χρόνια να περάσει κανεί τα σύνορα από τη Σλοβακία στην Αυστρία. Μια τραπεζική ή νομισματική ένωση θεωρείται ότι ήταν κάτι το απόλυτα μη ρεαλιστικό. Όπω είπε ο Νέλσον Μαντέλα, όλα φαίνονται ότι δεν είναι εφικτά μέχρι κάποιο να τα κάνει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θέλω μαζί σας και τα κρατη να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας που να βασίζεται σε πέντε πυλώνες. Πρώτα απ' όλα <clears throat> η ασφάλεια, η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κύρια αγορά ενέργειας με μισό δισεκατομμύριο καταναλωτές. 53% της ενέργειάς μας είναι εισαγόμενη σε κόστος 400 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Είμαστε ο μεγαλύτερος ενεργειακός πελάτης στον χρόνο, στον πλανήτη μας. Το δείχνουμε όμως αυτό. Έχουμε την ικανότητα να πιέσουμε για να έχουμε δίκαια αντίτιμα για την ενέργεια και καλύτερες συνδικές αγορές. Σίγουρα όχι. Η έλλειψη ικανότητά μα να έχουμε μια ενωμένη φωνή για τα θέματα αυτά περιορίζει την επιρροή μα. Πρέπει να είναι πιο αποφασιστική η ενεργειακή διπλωματία τη Ευρώπη, γιατί τα ενεργειακά μα συμφέροντα θα πρέπει να είναι μία από τι μεγαλύτερε προτεραιότητέ μα σε επίπεδο εξωτερικού εμπόριου και εξωτερική πολιτική. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στι πιέσει από τρίτε χώρε και να αποφύγουμε τι τρευλώσει αγορά από τρίτε χώρε που δεν σέβονται του κανόνε ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ υποστηρίζω μια ευρωπαϊκή συζήτηση που θα οδηγήσει σε μια συνένεση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να διαπραγματευτεί διεθνεί συμφωνίε εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε. Η δημιουργία τη Ενεργειακή Ένωση σημαίνει επίση καλύτερη συνεργασία με του γειτονέ μα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των αγορών Θέλω να τονίσω λοιπόν τη σημασία τη ενεργειακή κοινότητα για τα θέματα αυτά. Πρέπει επίση να διερευνήσουμε κοινού τρόπου αγορά φυσικού αερίου. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε του κανόνε ανταγωνισμού, του κανόνε του ΠΟΕ, αλλά θα πρέπει πιστεύω να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το γεγονό ότι αγοράζει ενέργεια 400 δισεκατομμυρίων ως ένα πιο ισχυρό επιχείρημα. Ο πραγματικός συντονισμός σημαίνει ότι κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να αλλάζει το ενεργειακό του μείγμα χωρίς να έχει συντονισμό με τους γείτονές του και χωρίς να καταλάβει τις συνέπειες για τους γείτονες αυτού αυτούς. Ένα περαιτέρω στοιχείο είναι η διαφοροποίηση της παροχής ε, ενέργειας σε ό,τι αφορά και τις διαδρομές και τους παρόχους ενέργειας. Θα πρέπει να εργαστούμε για τον νότιο διάδρομο για να έρθει φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με την ε, Νορβηγία, να προωθήσουμε ένα κεντρικό ε, ένα κέντρο ενέργειας για την Μεσόγειο αυτό συμπεριλαμβάνει καλύτερη συνεργασία με την Αλγερία και δημιουργία τερματικών σταθμών για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Επίση, πρέπει να έχουμε μια ανταγωνιστική και πλήρη εσωτερική αγορά. Μια πλήρη εσωτερική αγορά θα γίνει η ραχοκοκαλιά τη νέα Ενεργειακή Ένωση για την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει να αυξήσουμε τι διαμεθοριακέ ροέ ενέργεια, να έχουμε μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία και μια καλύτερα συνδεδεμένη υποδομή. Θα πρέπει να βελτιώσουμε εδώ την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, να την ενισχύσουμε και να την εφαρμόσουμε πλήρω για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να έχουμε προσιτέ τιμέ ενέργεια για τα νοικοκυριά, ιδίω για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Χρειαζόμαστε τη σωστή υποδομή για τα θέματα ενέργεια με σωστέ διασυνδέσει, ιδίω για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια στο δίκτυο ενέργεια και να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τι νησίδε ενέργεια. Χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα διορθωτικά ταμεία, το Connecting Europe Facility, τι κοινέ επενδύσει και το μελλοντικό πακέτο επενδύσεων Juncker, ώστε να ενισχύσουμε τα σχέδια αυτά υποδομών. Τρίτο, πρέπει να μπορέσουμε να περιορίσουμε την ζήτηση ενέργειας για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας και να βελτιώσουμε την ασφάλεια ενέργειας πρέπει να μειώσουμε την συνολική ζήτηση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ο πρώτος, ο πιο εύκολος πόρος ενέργειας. Το καλύτερο μεγαβάτ είναι ένα μεγαβάτ που δεν καταναλώνεται ποτέ. Η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά επέκεινα του 2020. Η βελτίωση της αποδοτικότητας δεν θα αυξήσει μονάχα την ενεργειακή ασφάλεια, θα δώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πλήρως υποστηρίζω την δέσμευση του κυρίου Γιούνκερ για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και τονίζω ότι η υποτεραιότητά μας θα πρέπει να τα κτίρια, οι μεταφορές και η παραγωγή προϊόντων τέταρτο στοιχείο είναι η μείωση του περιεχομένου άνθρακα στην παραγωγή ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να μειώσουμε τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για του στόχου μα του 2030 και είμαι απόλυτα προσιλωμένο στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη αγορά για τα θέματα ανανεώσιμων ενεργειών. Ήδη το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγή 44% ηλεκτρισμού από ανανεώσιμη ενέργεια. Είμαστε πρώτοι και στι τεχνολογίε ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία μα και για τη δημιουργία πάνω από 4, 4 εκατομμυρίων πρασίνων θέσεων εργασία. Φυσικά τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα να έχουν το δικό του μείγμα ενέργεια, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια κοινή συμφωνία το 2015 στο Παρίσι για του στόχου αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει παίξει πρωτοπόρο ρόλο θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο. Το τελευταίο στοιχείο, πέμπτο πυλώνα, είναι η έρευνα και η καινοτομία. Χρειάζονται περαιτέρω επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία και είναι κεφαλαιώδη, ιδίω για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τι τεχνολογίε τη να φέρει αυτές τις τεχνολογίες της χαμηλού κόστους και χαμηλής χρήσης άνθρακα, υψηλής απόδοση τεχνολογίας στην αγορά. Αυτές οι τεχνολογίες είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 για κλιματική αλλαγή, για ενέργεια, οικονομικά και κοινωνικά θέματα και περαιτέρω. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα πέντε, αυτά τα πέντε βασικά στοιχεία, οι πέντε πυλώνες επί των οποίων μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση η οποία να βασίζεται με μια προορατική πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ του. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα και όχι το άλλο. Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκομίσει καρπού και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο περιβάλλοντο και να δημιουργήσει τι θέσει εργασία που θα δώσει πράσινη ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Πριν από δύο εβδομάδε ήμουνα ενώπιον ε, τη Επιτροπή Μεταφορών για την ακρόασή μου για τι μεταφορέ και τα θέματα διαστήματο. Σήμερα προσπαθώ να κερδίσω την υποστήριξή σα για το νέο χαρτοφυλάκιο το οποίο μου δόθηκε την προηγούμενη Τετάρτη. Δεν ισχυρίζομαι ότι έγινα από τη μια μέρα στην άλλη εμπειρογνώμο στα θέματα ενέργεια. Έκανα όμω ό,τι μπορούσα για να προετοιμαστώ όσο μπορούσα καλύτερα για αυτή την ακρόαση. Και αν έχω την υποστήριξή σα, θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε από κοινού την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μάθω όλα αυτά που χρειάζονται για αυτά. Γιατί πιστεύω πολλά μπορούν να γίνουν σε πέντε χρόνια. Πιστεύω ότι όλοι μας το οφείλουμε στους πολίτες για να εξασφαλίσουμε ότι το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Τώρα είναι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε και τώρα θα περάσουμε στον πρώτο γύρο παρατηρήσεων και ερωτήσεων εκ μέρους των πολιτικών ομάδων καταρχήν. Ο κύριος Κρυσιάννη Κάριμς εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεύκοβιτς. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι θα πρέπει να σημαίνει να εξηγηθεί κανεί εντό πέντε ημερών με ένα εντελώ νέο χαρτοφυλόκιο. Νομίζω ότι όλοι εδώ κατανοούμε την κατάσταση στην οποία βρεθήκατε. Ωστόσο, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ασφάλεια του εφοδιασμού. Όπως ε, ξέρετε και όπως είπατε, εμείς εξαρτώμαθα πάρα πολύ στις εισαγωγές ενέργειας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τη μέρα. Και ο τομέας του αερίου θέτει πάρα πολλές ε, προκλήσεις γιατί είναι δύσκολη η μεταφορά μέσω αγωγών. Επίσης, στον τομέα του αερίου έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από την παροχή από την αερίου από τη Ρωσία. Και εσείς ο ίδιος αναφέρατε ότι ε, η, στην Ουκρανία, η χρησιμοποιείται σαν ε, όπλο. Δύο ερωτήσεις. Εσείς ως ε, Επίτροπος θα υποστηρίξετε τον αγωγό South Stream ο οποίος θα αυξήσει την ανεξαρτησία από την Ρωσία και δεύτερον πώς προτείνετε να μειωθεί η εξάρτησή μας από την Ρωσία και να αυξηθεί συνολικά η ασφάλεια εφοδιασμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο ερωτήσεις που είναι απολύτως ε, ε, σημαντικές και θα καθορίσουν το έργο μου τα προσεχή πέντε χρόνια. Θα αναφερθώ καταρχήν στο South ε, Stream, το οποίο, το οποίο η λειτουργία έχει ανασταλεί. Και επειδή δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα τόσο μεγάλο έργο να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας εταιρεία η οποία δεν σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε δύο βασικές ερωτήσεις που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Πρώτον, μια απόλυτη προσήλωση προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεύτερον αυτό το οποίο περιγράφεται πολύ καλά στο, στη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ενέργεια και Ασφάλεια πώς αυτό θα βοηθήσει την άξιο επίπεδα ασφάλεια στην Ευρώπη, πώς δηλαδή θα διαφοροποιηθούν οι πηγές μας ενέργειες. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ε, βλέπω το εγχείρημα αυτό πραγματικά να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό πιστεύω ότι μελλοντικά θα στρέψουμε ε, τις προσπάθειές μας και τις επενδύσεις μας προς τον νότιο διάδρομο. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί θα μας βοηθήσει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ενέργειας, να πάρουμε αέριο από την Κασπία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε τη δυνατότητα να μην περιοριζόμαστε στις πηγές ε, του Αζερβαϊτζάν, φυσικού αερίου, αλλά να αναπτύξουμε μια καλή συνεργασία, ούτε ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και με άλλη σημαντική πηγή, ε, το Τουρκμανιστάν. Η ξεκάθαρη προτίμησή μου λοιπόν να υπάρξει μια διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τα έργα για τον νότιο διάδρομο να εξελιχθούν και να τα υποστηρίξουμε πολιτικά πλήρως. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των σοσιαλιστών η κυρία Καθλίν Βαν Μπέμπτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε έχω κρυώσει και η φωνή μου είναι λίγο βραχνή. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι για την Ενεργειακή Ένωση του σύνολό τη. Όπω ξέρετε, υπάρχουν ήδη διάφορε ερμηνείε και ε, ε, σε σχέση με την προσπάθεια να γίνουμε ανεξάρτητα από τη Ρωσία. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για τη δική μας ομάδα. Εσείς αναφέρατε πέντε συγκεκριμένους πυλώνες που νομίζω καλύπτουν ε, την πλειονότητα αυτού που ονομάζουμε Ενεργειακή Ένωση. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο βασικές ερωτήσεις. Εάν δούμε αυτούς τους πέντε πυλώνες, ποιες, θα είναι, είναι οι δικές σας βασικές προτεραιότητες και ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα παίρνετε εσείς για τα προσεχή έτη. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Πιστεύω ότι βεβαίως οι από αυτέ τι προτεραιότητε μπορούμε να προγραμματίσουμε και να συνεργαστούμε και ε, νομίζω ότι ορισμένε αυτές θα πάρουν σάρκα και οστά. Ε, θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αύριο που θα έχει ο αντιπρόεδρος κ. και η Ρώση και η Ουκρανία. εταίροι. Ελπίζουμε να βρεθεί μια συμφωνία και να αποφύγουμε μια δραματική κατάσταση όσον αφορά την παροχή αερίου το χειμώνα στην Ουκρανία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, ανησυχώ βεβαίως ε, ε, για το θέμα αυτό και αυτή είναι η άμεση μας προτεραιότητα. Αλλά εάν βάλουμε αυτό παράμερα, εάν ε, δούμε τι γίνεται από στρατηγική άποψη, νομίζω ότι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση θα ήταν να προωθήσουμε όλους τους πυλώνες από κοινού. Γιατί υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ε, ταυτόχρονα και ελπίζω ότι θα έχουμε γρήγορα φιλόδοξε αποφάσεις του Συμβουλίου. Αύριο θα εκπροσωπήσω την Επιτροπή στο Συμβούλιο και πραγματικά αναμένω πραγματικά ε, θετικά αποτελέσματα ε, και την προετοιμασία των Ευρωπαίων, ε, τη συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα μεταφέρουμε αυτό το πακέτο στο νομικό πλαίσιο, στο νομοθετικό πλαίσιο. Και την άνοιξη θα προετοιμάσουμε τη δική μας ε, θέση για ε, το Παρίσι. Και βεβαίως... Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τα προγράμματα όσον αφορά το εργαλείο για τη διασύνδεση της Ευρώπης και να υπάρξει μια σωστή διαδικασία επιλογής και διαγωνισμών, ε, προκήρυξης διαγωνισμών για το καλύτερο πρόγραμμα. Ε, θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα της εσωτερικής αγοράς, γιατί ξέρετε ότι ήδη έχουμε συμφωνήσει ότι το 2014 θα έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη και γνωρίζετε το αποτέλεσμα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο τέλος αυτού του χρόνου. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχαίως. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζούλη Γκέρλινγκ έχει το λόγο από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Καλώς ήρθατε κύριε Σεύκοβιτς. Μέσα στη δομή που έχει δημιουργήσει ο κύριος Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος για την ενέργεια παίζει ένα κομβικό ρόλο για να μπορέσει να επιβλέπει το έργο των επιτρόπων στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Αλλά μέχρι στιγμής οι αντιπρόεδροι δεν έχουν δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφή σε σχέση με τον ρόλο τους. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή Τώρα, σε σχέση με την ε, παρακολούθηση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε από τη μια μεριά τα θέματα στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή που περιλαμβάνουν τα αέρια θερμοκήπιων, ενώ τα, οι άλλε εκπομπέ δεν λαμβάνουν υπόψη σε αυτό το πακέτο. Δεν υπάρχει συνέργεια, δεν συμπληρώνονται μεταξύ του αυτά τα δύο εγχειρήματα και οι ημερομηνίε δεν ταιριάζουν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν εκτικούς στόχους. Δεν είναι αυτή η καλύτερη νομοθεσία λοιπόν και πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρλινγκ. Παρουσιάστε μια κατάσταση που δεν ήταν και η βελτιότερη και γι' αυτό ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν θέλησε να αλλάξει η δομή της Κομισιόν γιατί αυτό θα δημιουργήσει δυνατότητα συνεργασία από την αρχή όλων των εγχειρημάτων, όχι μόνο για τους επιτρόπους αλλά και για τις υπηρεσίες τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αρμόδιος ε, αντιπρόεδρος και οι αρμόδιοι επίτροποι να μπορέσουν να δώσουν το σωστό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ τους. Αν δείτε το νέο οργανόγραμμα της Κομισιόν, αυτή είναι η θέση που θα έχω αν με εγκρίνετε μετά από αυτή την ακρόαση και αυτοί είναι οι επίτροποι τους οποίους πρέπει να συνδενήσω. Σας τονίζω εδώ πέρα ότι το χρώμα που με αντιπροσωπεύει εδώ είναι πράσινο. Θα είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστώ στενά με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μπορώ λοιπόν να σας υποσχεθώ ότι από τη δική μου οπτική γωνία ο ρόλος του Αντιπροέδρου είναι ρόλος συντονιστή είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εξασφαλίσει ότι συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες από την αρχή και έτσι δεν θα έχουμε μια υπηρεσία να ζητάει ένα σύνολο στόχων ενώ μια άλλη υπηρεσία έχει διαφορετικούς στόχους ή έχουν διαφορετικά συστήματα για να παρέχουν αναφορές η κάθε υπηρεσία. Και έτσι όταν φτάνουμε στο καταληκτικό στάδιο, στο σώμα των επιτρόπων, δεν θα υπάρχουν προβλήματα συγκρούσεων γιατί το, το γραφείο κάθε επιτρόπου προσπαθεί να φέρει τα πράγματα προς τη μια ή προς την άλλη μεριά. Είναι δύσκολο λοιπόν στο τελικό στάδιο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Θέλουμε να αναστρέψουμε αυτή τη λογική, θέλουμε από την αρχή να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι προχωρούμε από κοινού και να εξασφαλίσουμε επίσης ότι δεν θα χρειάζεται να υπάρχει τη γραφειοκρατία και παράδοση εκθέσεων και υπερβολικές υποχρεώσεις για εκθέσεις όπως το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Φέντερ λέει <clears throat> από την ε, φιλελεύθερη ομάδα είναι και αντιπρόεδρο μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Εδώ είμαι. Έχω πάρει νέα γραφεία στο γραφείο μου ώστε όταν ξανάρθετε να με επισκεφτείτε θα είσαστε πιο άνετα. Εσείς ουσιαστικά έχετε απαντήσει στο πρώτο ερώτημά μου που είναι πώς θα μπορέσετε να γίνετε μια πρωτοπόρα να γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρα δύναμη στι ανανεώσιμε ενέργειε. Υπάρχει συνεχή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη γεωπολιτική, για την οικονομική ανάπτυξη και για την ανανεώσιμη ενέργεια. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα πούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αναχαιτίζεται από την ανάγκη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να πείτε λίγο περισσότερα για το θέμα αυτό. Βλέπετε την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να απειλεί την οικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση. Πιστεύω ότι και η βιομηχανία η βιομηχανική ανάπτυξη και μια ανταγωνιστική πολιτική για την πράσινη οικονομία πρέπει να αλληλοϊποστηρίζονται. Εσείς είσαστε στις επιτροπές σας οι αρμόδιοι για τα θέματα περιβάλλοντος ενέργειας και ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το τίμημα των εισαγωγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η αστάθεια που αντιμετωπίσουμε και αυτό γίνεται ουσιαστικά κάθε φθινόπωρο. Αναδύεται πάλι αυτό το πρόβλημα γιατί εξαρτώμαστε πάρα πολύ από ενεργειακές πηγές έξω, της, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι. Οι εναλλακτικέ ενέργειες μας δίνουν λοιπόν εγχώρια ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο η ηλιακή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια κτλ. Όλα αυτά μπορούμε να τα έχουμε στην Ευρώπη και οι εταιρείε μας είναι οι πρωτοπόροι σε παγκόσμιο επίπεδο για τις τεχνολογίες αυτές ανανεώσιμων ενεργειών και είναι πάρα πολύ επιτυχημένες και σε άλλες αγορές, σε χώρες όπως είναι η Κίνα όπου αρχίσουν να καταλαβαίνουν και εκεί οι πολίτες ότι δεν έχει νόημα να τρέξει μαραθώνιο φορώντας μια μάσκα επειδή είναι μολυσμένη η ατμόσφαιρα και δεν έχει νόημα να κλείνεται βιομηχανίες για να μπορούν να βλέπουν οι θεατές στους Ολυμπιακούς Αγώνες ποιος τρέχει σε ποια διαδρομή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε μια πρόοδο και θα δώσουμε ένα σωστό πλαίσιο και ένα καθεστώς νομικής ασφάλειας στις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, ώστε να προωθήσουμε τις πράσινες τεχνολογίες με έναν τρόπο ο οποίος δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά δίνει προσιτή και καθαρή ενέργεια, πράσινη ενέργεια, η οποία θα βοηθήσει και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Σιλικιώτης από την ΚΟΕ. Κύριε Αντιπρόεδρε, στην ανακοίνωση της Κομισιόν με θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναφορά στα μεγάλα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας ούτε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση κύριε Σεύκοβης αναβερθήκετε σε αυτά ε, τα κοιτάσματα ε, αναφέρεστε μόνο γενικά στη δημιουργία ενός μοσιακού κόμβου. Ε, πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν αυτά τα κοιτάσματα και ιδιαίτερα τα κοιτάσματα που ανεβρέθηκα στην Κύπρο να πω ότι τώρα ε, προχωρούν ε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε σημαντικές φιλόδοξες ερευνητικές γεωτρήσεις. Είναι στις προτεραιότητες σας ακριβώς να αναπτυχθεί ένας μεσογειακός κόμβος μέσω διαδρόμου από την νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί έναν έργο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε αυτήν την περιοχή. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα πράγμα το οποίο αναφέρθηκε στις ε, πρώτες μου παρατηρήσεις αλλά με την πίεση του χρόνου δεν μπορούσα να τα πω όλα. Εγώ αναφέρθηκα ε, στον Μεσογειακό κόμβο, ενεργειακό κόμβο. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει το κοίτασμα της Αφροδίτης, είναι νέα οικόπεδα τα οποία έχουν, έχουν τη δυνατότητα μεγάλης παραγωγής όσον αφορά το αέριο, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη έρευνα και ενδεχομένως να βρεθούν μεγαλύτερα αποθέματα. Ε, ε, υπάρχουν βεβαίως προβλήματα για χώρες, δύσκολη κατάσταση για χώρες όπως ε, η Κύπρος ή η Μάλτα έτσι ώστε να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα που έχουν ως νησίδες ενέργειας. Θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη η οποία να ξεπερασουν αυτο το προβλημα που εχουν ως νησιδες ενεργειας θα πρεπει να δειξουμε λιγη η οποια να φανει και στον κατάλογο των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά το ξεκλείδωμα αυτών των νησίδων αλυσίδων ενέργειας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται και θα συνεργαστεί με την ε, ε, Κυπριακή κυβέρνηση έτσι ώστε να ερευνηθεί περαιτέρω το οικόπεδο Αφροδίτη και να βεβαιωθούμε ότι η Κύπρος θα συνδεθεί με τον, με τον ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης και θα περιμένουμε καινούριε αποκαλύψεις, ανακαλύψεις και ε, καινούρια μεγαλύτερη συμμετοχή και της Κύπρου ε, σε αυτήν την μικρότερη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικές πηγές. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εγώ εδώ είμαι κύριε Σαφκοβίτσα. Ε, όσον αφορά τις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις ε, για το κλίμα. Ε, παραμένει ασαφές ένα συγκεκριμένο απλό ερώτημα. Ποιος θα διαπραγματευτεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ένα όνομα χρειαζόμαστε έτσι ώστε να ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, όσον αφορά το περιεχόμενο, είπατε επανειλημμένα ότι θέλετε να είναι ουσιώδης η ε, ε, διεθνής εξέλιξη. Τι εννοείται ουσιώδης. Ε, τι, σημαίνει για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει ένα, ε, ε, θέλει, έχει πιθανότητα 40% ε, έτσι ώστε να επιτύχει το, το στόχο της. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν και οι υπόλοιπε συνθήκες είναι αυτές και έτσι ώστε να ξέρουμε ότι το μείον 40 είναι όντως μείον 40 και όχι μείον 50. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, εάν το πρόβλημα είναι ποιο θα πάει στο Παρίσι, εγώ θα πάω στο Παρίσι αλλά είναι μακρύς ο δρόμος που οδηγεί στο Παρίσι ε, και ξεκινάει ήδη από την Τρίτη στις Βρυξέλλες και μετά θα συνεχιστεί στη Λίμα και μετά θα υπάρξουν και άλλες πολλές διεθνείς διασκέψεις και συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει κανείς ε, είναι ε, να δείξει αποφασιστικότητα και ε, πνεύμα ρωμαλαίων. Γιατί το θέμα δεν αφορά μονάχα τον Αντιπρόεδρο για την Ένωση της Ενέργειας, αλλά όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που σας έδειξε προηγουμένως στο οργανόγραμμα είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τα οποία συνδέονται και με την Ενεργειακή Ένωση αλλά και με την ε, εν τέλει επιτυχία στο Παρίσι. Αυτό που θα ήταν το πιο αποτελεσματικό και η καλύτερη αντιπροσώπευση στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι ε, η καλή εκπροσώπηση της ε, Κομισιόν και αυτό δεν αφορά μονάχα το αν θα πάει ο αντιπρόεδρος ο οποίος ασχολείται με θέματα ενεργειακής ένωσης. Το θέμα είναι να έχουμε επιτυχία, να επιτύχουμε διεθνή νομικά δεσμευτική συμφωνία στο Παρίσι γιατί το κλίμα είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και πρέπει ε, να είμαστε σίγουροι ότι και οι πολίτες θα είναι ικανοποιημένοι αλλά και η βιομηχανία δεν θα οπισθοδρομήσει. Ε, όσον αφορά το επίπεδο των ε, ε, φιλοδοξιών, οπωσδήποτε την Τρίτη θα ξέρουμε κάτι παραπάνω μετά από την έγκριση του πλαισίου για το 2030. Ωστόσο, σας λέω από τώρα ότι η προετοιμασία της Κομισιόν θα είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά το Παρίσι. Ευχαριστώ θα ολοκληρώσαμε τον ε, κύκλο των, πολιτικών, των εκπροσώπων των πολιτικών ε, ομάδων. Ο συνάδελφος Πίτερ Λίζε τώρα. Ναι κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, κύριε πρόεδρε, αναφερθήκατε στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και ο Μικέλ Αρίας Κανιέτε ήταν πολύ ακριβείς ως προς το ερώτημα αυτό. Δηλαδή 30% ε, δέσμευσης μέχρι το 2030 και θα ήθελα να μου το πείτε και εσείς με ακρίβεια και το πώς ε, μπορείτε πραγματικά να υποστηρίξετε αυτούς τους δύο να εφαρμόσουν αυτή τη δέσμευση. Το θέμα των κονδυλίων είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει η οδηγία Eco Design ε, και ε, παρόλο που είναι λογική προς τον πυρήνα της, ωστόσο έχουν εκφραστεί και κάποιες ε, κριτικές. Ε, ε, ερώτημα, τι θεωρείτε για την ρύθμιση των ντους όσον αφορά την οδηγία είπε ο κύριος Κανιέτε ότι θέλει να την συνεχίσει. Αλλά πώς ε, θέλετε εσείς να αφαιρέσετε το κομμάτι της ε, γραφειοκρατίας και να δώσετε ρεθίσματα ούτως ώστε να υπάρξει υποστήριξη. Thank you, thank ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Λίζε ε, ε, βεβαίως όπως είπε ο, ο πρόεδρος κ. Ε, Γιούγκερ και ο συνάδελφος Μικέλ και εγώ έχω αναλάβει τη δέσμευση του 25% στον πρώτη ενεργειακή αποδοτικότητα και θα κάνω ό,τι μπορώ ήδη αύριο στο Λουξεμβούργο. Και μπορώ να σας πω ότι όταν προετοιμαζόμουν για τη σημερινή ακρόαση αλλά και για τις αυριανές διαπραγματεύσεις με τους ε, υπουργούς, ε, τα θέματα αυτά θα είναι εξαιρετικά δύσκολα στη διαπραγμάτευση ε, γιατί θα υπάρξει μεγάλη αντίσταση αντιπολίτευση από τις χώρες μέλη. Αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά στην πραγματεύσεις αύριο για να εξηγήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η στόχη για το μέλλον ε, της πράσινης πολιτικής στην Ευρώπη. Όσον αφορά το eco-design, εδώ ε, νομίζω ότι η Επιτροπή, το σύνολο της Επιτροπής θα χρειαζόταν τη βοήθειά σας όσον αφορά μια καλύτερη επικοινωνία. η οδηγία αυτή ε, έχει περιγραφεί στον τύπο και περιγράφεται σαν ένα γραφειοκρατικό εργαλείο μέσω της οποίας η Επιτροπή προτίθεται να ρυθμίσει τα πάντα από τις μικρές στις μεγάλες αφαρμογές. Και λησμονούμε να πούμε ότι χάρη σε αυτή την οδηγία το 2020 η Ευρώπη πρόκειται να εξοικονομήσει ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί την ε, κατανάλωση ενέργεια στην Ιταλία για ένα χρόνο. Τόσο σημαντικό είναι αυτό ο στόχο, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει απλώ να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία προ τα έξω. Ε, όσον αφορά τις ηλεκτρικές σκούπες, προτάσει όπω αυτή θα πρέπει να εξηγήσουμε στου πολίτε γιατί το προτείνουμε, ποια θα είναι τα συγκεκριμένα ωφέλη και να αποφύγουμε αυτή τη γραφειοκρατία στην οποία αναφερθήκατε. Και συμφωνώ μαζί σα, θα πρέπει να μειωθεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνες τις εφαρμογές που πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Ματίας Κρότε. Ευχαριστώ πολύ εδώ είμαι. Όταν πήραμε τα χαρτοφυλάκια για την Επιτροπή και ανακαλύψαμε εκεί το θέμα της Ενεργειακής Ένωσης και το γεγονός ότι το κλίμα συνδέεται με την ενέργεια ε, υπήρξαν πολλές επιφυλάξεις από τους συναδέλφους ότι τα επόμενα πέντε χρόνια το θέμα της κλιματικής πολιτικής αλλά και το θέμα της περιβαλλοντικής πολιτικής τελικά ε, θα μπει στην ε, άκρη, θα παραμεληθεί. Ε, τι σκέφτεστε εσείς ως αντιπρόεδρος να κάνετε για αυτό το τομέα γιατί οι φωνές της ε, κριτικής ε, μετριάζονται ε, αναφερθήκατε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είπατε κάποια συγκεκριμένα πράγματα αλλά τι πιστεύετε για το θέμα αυτό και σε σχέση με την κοινή γνώμη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ υπογραφές από πολίτες. Τι θα γίνει με το περιβάλλον, αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρότε για αυτό το ερώτημα. Ε, καταρχήν δεν ε, πιστεύω ότι αυτή η πολύ σημαντική περιβαλλοντική πολιτική θα μπει στην άκρη. Γιατί ε, ε βεβαίω ξέρω πώς σας ενδιαφέρουν οι πολιτικές αυτές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και αυτό αναγράφεται και στο Mission Letter ε, ε, σε, μένα στον, ε, προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρονται οι στόχοι αυτοί, οι προτεραιότητες αυτές και αναφέρεται πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές αυτές για το μέλλον. Βεβαίως θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, ε, υπάρχει τρίτη... Υπάρχει τρίτη, μια τρίτη πηγή παραγωγής ενέργειας. Αλλά πολύ συχνά η ευρεία χρήση ενέργειας ε, ε, είναι περιορισμένη γιατί δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται αυτή η μορφή ενέργειας ε, και υπάρχουν πολλά εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο του, της ηλεκτρικής ενέργειας. Και βεβαίως ε, θα θέλαμε να υπάρξει περισσότερη έρευνα και περισσότερα αποτελέσματα ερευνητικά, ούτως ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των πηγών αυτών. Ε, και ξεκάθαρα αυτή θα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής γιατί όταν μιλούμε για αυτόχθονες ε, πηγές ή για ανεργιακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, αυτάρκεια μάλλον, ή για τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε ως ε, ανεπτυγμένο μέρος ε, αυτού του κόσμου ως προς το 2015 τα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο παράγον κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ. Ο Άιαν Ντόγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ στα θέματα της ενεργειακής υποδομής. Περιμένετε να υπάρξει ανάγκη για μια νέα συνθήκη ή κάποια αλλαγή των συνδικών για να μπορέσει να υπάρξει ένα ισόπεδο γήπεδο ανταγωνισμού για τα θέματα ε, υποδομών ενέργειας. Ως ε, σκότος ε, ευρωβουλευτής πρέπει να σας πω ότι η Σκοτία έχει πολλές πηγές ενέργειας αλλά δεν είναι καλά διασυνδεδεμένη. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την αιωλική ενέργεια εάν δεν είναι πραγματικά διασυνδεδεμένος σε ένα δίκτυο. Πόσο, κονδύλια λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε, θα προσδιορίσετε ακριβώς για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου και θα ήθελε ο λαός της Σκοτίας να ξέρει πολύ καλά αν αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες σύνδεσης για τα ενεργειακά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σεύτσοβιτς. Πιστεύω ειλικρινά ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με την τωρινή συνθήκη ήδη. Ξέρετε ότι είναι ακόμα πολύπλοκο το να αλλάξει η συνθήκη. Θυμόσαστε ότι η Επιτροπή Μπαρόσο 2 καθυστέρησε να αναλάβει το έργο της λόγω της διαδικασίας κύρωσης των συνθήκων. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν λοιπόν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να εξαντλήσουμε καταρχήν το περιθώριο που έχουμε σε πολιτικό και νομικό επίπεδο με την τωρινή συνθήκη εγώ πιστεύω μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα υποδομών και τις διασυνδέσεις των ενεργειακών δικτύων. Έχουμε πολλές δυνατότητες για τη χρηματοδότησή τους. Η πρώτη δυνατότητα είναι βέβαια η διευκόλυνση Connecting Europe, Connecting Europe Facility, η οποία χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό σε επίπεδο 6 δισεκατομμύριων ευρώ περίπου. Δεν είναι τεράστιο αυτό το ποσό. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμε και δημιουργικές τεχνικές χρηματοδότησης. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνικές για να δημιουργηθούν για να φτάσουμε στα 300 δισεκατομμύρια επενδύσεων που, αν, που ανήγγειλε ο πρόεδρος Ιούνκερ. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Για μένα αυτό που είναι θετικό είναι ότι έχουμε ένα γενικό κατευθυντήριο σχέδιο για το πώς θα πετύχουμε τους ενεργειακούς μας στόχους. Έχουμε λοιπόν ένα παράτημα της στρατηγικής που αναφέρει τους συγκεκριμένους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατό. Τα συγκεκριμένα ενεργειακά σχέδια πρέπει να περατωθούν το ταχύτερο δυνατό και αυτά που πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο μέσο πρόθεσμα. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν με την σωστή δημιουργία αυτού του πακέτου επενδύσεων, μπορούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προχωρήσουμε και πέραν αυτού του πακέτου για να χρηματοδοτήσουμε μελλοντικέ υποδομέ ενέργεια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Μπούσεκ. Ο κύριο Χερμπράντι έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. <clears throat> Εδώ στο κέντρο είμαι. Κύριε Σεύτσοβιτ, σα ευχαριστώ. Αναφερθήκατε για τους πέντε πυλώνες σας, στους πέντε πυλώνες την ενεργειακή απόδοση και την μείωση της χρήσης άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας, βλέπω ότι στις απαντήσεις σας εσείς εστιάζετε πάρα πολύ στα ορυκτά καύσιμα και την ασφάλεια εφοδιασμού. Θα συμφωνούσατε όμως μαζί μου ότι το να είναι λιγότερο πολυδάπανη, λιγότερο βρώμικη η ενέργεια στην Ευρώπη και να εξαρτώμαστε λιγότερο από τις εξωτερικές πηγές θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις ανανεώσιμες ενέργειες και η Ανατολική Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει για να πετύχει το στον αυτό περισσότερο στην, στις ανανεώσιμες ενέργειες. Τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαίρεση μεταξύ Ανατολή και Δύσης στο Συμβούλιο. Θα μπορέσετε να πείσετε του εταίρους μα από την Ανατολική Ευρώπη ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ενεργειακή και κλιματική πολιτική γιατί αυτό είναι προ το δικό του συμφέρον ήδη. Σα ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και σίγουρα θα κάνω ήδη αύριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ό,τι περνάει από το χέρι μου για το στόχο αυτό. Για μένα το πιο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης είναι να μπορέσουμε να έχουμε σαφείς ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκές συμφωνίες για τα θέματα αυτά, να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη κινείται όλη προς μία κατεύθυνση, έχει μία ενιαία αντιμετώπιση και έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για να πετύχουμε όχι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα μέχρι την συνδιάσκεψη του Παρισιού του χρόνου, αλλά μέχρι το 2020, 30 και 50. Αν δούμε τους στόχους που έχουν θεσπιστεί για το 20, για το 2030 η Κομισιόν κάνει σαφείς αναλύσεις αντικτύπου επί τη βάση της δέσμευσή μας ότι μέχρι το 2005 ο ανεπτυγμένος κόσμος θα πρέπει να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 ή 90%. Με αυτό το σημείο εκκίνησης καταλήγουμε στα στοιχεία τα αριθμητικά τα οποία προτείνουμε σε εσά και στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι όλο και περισσότερο σαφές και στις χώρες κεντροανατολικής Ευρώπης ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια. Υπάρχει πρόοδος, ακόμα βέβαια έχουμε διαφορετικά σημεία κίνησης για τις χώρες αυτές, διαφορετικές δυνατότητες χρηματοδότησης και διαφορετικές μορφές ε, δικτύων με διαφορετική ικανότητα να ενσωματώσουν την ανανεώσιμη ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε δύο στοιχεία στο πακέτο αυτό το οποίο θα συζητήθει την Πέμπτη. Πρώτον να έχουμε μία ε, θέση από κοινού και κατανομή προσπάθειας και δεύτερον αυτό το ταμείο επενδύσεων που θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ετήσια ε, χρηματοδότηση από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ώστε να μπορέσουν οι ενεργειακοί σταθμοί, η παραγωγή ενέργειας να ε, ανανεωθεί και να είναι πιο καθαρή και πιο αποδοτική από την σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις γραπτές σας απαντήσεις, κύριε Επιτροπέ, ε, ε, ε, είπατε ότι όλα τα κράτη-μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν πληροφορίες σωστές όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις και να καταλαβαίνουν ότι είναι ενωτική και ενιαία η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις πάλι σε διεθνές επίπεδο και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τις ε, εκπομπές, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, ε, και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν ε, μολυντές μεγάλοι, όπως είναι ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα. Τι μπορείτε να κάνετε για χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Μπορείτε να βελτιώσετε επίσης ε, την κατάσταση όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, έχω την ε, δυνατότητα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ε, μπορούμε οι δυο μας να συνενεθούμε ε, άνετα και οι διερμηνείς θα μεταφράσουν την απάντησή μου στα σλοβακικά. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας, μπορώ να σας υπασχεθώ εκ μέρους της Επιτροπής αλλά και σαν δική μου προσωπική δέσμευση ότι θα προετοιμάσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ότι θα έχουν ε, μεγάλο βαθμό, υψηλό βαθμό διαφάνειας και θα ενημερθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαπραγματευτικές θέσεις γιατί γνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο. Μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είμαι πολύ πιο αισιόδοξο όσον αφορά τους στόχους για το Παρίσι. Νομίζω ότι θα πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο Παρίσι από ό,τι είχαμε θεωρήσει αρχικά. Ε, στη Νέα Υόρκη ε, βιώσαμε κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή μια μεγαλύτερη δέσμευση για τους κλιματικούς στόχους και ε, Είδα ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μπαν Κιμούν, ε, πραγματικά είναι επίσης πρόθυμο να δεσμευτεί στην κατεύθυνση αυτή. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε ψήφισαν μια νέα νομοθεσία για του σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η Κίνα ε, αυτή τη στιγμή δοκιμάζει ένα καινούριο σύστημα το οποίο μοιάζει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας των ε, Ρήπων των εκπομπών αερίων και όλα αυτά προτίθεμα να τα αξιοποιήσω την Πέμπτη ούτω ώστε να ενισχύσω την ε, διαπραγματευτική μας ε, θέση για την άνοιξη του προσεχούς ε, έτους και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε περισσότερα ατού στα χέρια μας και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να λάβουν μέρος στα περισσότερα κράτη. Ο κύριος Γιάννη Γιάντος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε υποψήφι, εδώ βρίσκομαι, στα αριστερά σας. Μας είπατε και ε, άλλωστε αφορά και την ε, ε, επιστολή που περιγράφει την θέση σας του ε, ε, πρόεδρο Γιούγκερ ότι ε, θα επιτύχετε τους καλύτερους στόχους. Πιστεύετε όσον αφορά τις ανανεώσιμες, το 27% που έχει αναφέρει ως στόχο η παλαιά Επιτροπή και είσαστε μέλος του παλαιού ε, κολεγίου των Επιτρόπων και επομένως ψηφίσατε και εσείς τα μέτρα. Πιστεύετε ότι με το 27% η Ευρώπη θα, μειώσει τελικά κατά 50% την ικανότητά της όσον αφορά παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή θα γίνει με, λιγότερη ε, ε, προσπάθεια σε αυτή τη δεκαετία από τη δεκαετία 20-30. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ε, πρωταγωνιστής παριθμόν ένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απάντηση είναι θεμητή η ερώτησή σας. Θα σας εξηγήσω ποια είναι, αυτή, ποια είναι η λογική της προτάσεως που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σημείο κίνηση στην αρχή ήταν πώς μπορούμε να καλύψουμε τις δεσμεύσεις μας ε, ε, όσον αφορά τον στόχο της μείωσης ε, της χρήσης άνθρακα για το 2030 και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον πιο λογικό από οικονομικής απόψεως τρόπο. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το σημείο κίνηση της ανάλυσης και προσπαθήσαμε να βρούμε μεθοδολογικά πώς μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Ε, ε, λάβαμε υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους τις οποίες σας παρουσίασα ε, και που τα κράτη-μέλη συμφώνησαν με αυτό το μείον 40 όσον αφορά την μία των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και είπαμε τουλάχιστον 27% όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί αυτό θα ήταν ο πιο σωστός από απόψη απόδοσης τρόπος. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πιο γρήγορα αλλά το κόστος θα ήταν πάρα πολύ ψηλότερο και επομένως κάναμε και μία οικονομική ανάλυση ταυτόχρονα έτσι ώστε ε, να προτείνουμε κάτι και σε εσά και στα κράτη-μέλη που θα ήταν πιο λογικό από οικονομική απόψεως. Μπορώ να σας πω ότι ήδη τώρα είμαι πεπισμένος ότι θα ε, ξεπεράσουμε αυτό το στόχο του 27% γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες είναι διατεθειμένες να ξεπεράσουν αυτό το στόχο του 27%. Πιστεύω δε ότι και κατά την άποψη αυτή τελικά ε, η Ευρώπη θα ε, επιτύχει τον στόχο αυτό και θα τον ξεπεράσει. Και αυτό προς όφελος ε, των προσπαθειών μας για την κλιματική αλλαγή και κυρίως όσον αφορά τον στόχο για την μείωση άνθρακα. Jean-Luc Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα σας υπογραμμίσατε τις, οικονο, ε, τις οικονομίες ενέργειας, αναφερθήκατε ε, στα 300 δις ε, τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος Γιούγκερ και τα υποσχέθηκε σε πολλούς επιτρόπους χωρίς να ξέρουμε όμως αν υπάρχουν αυτά τα 300 δις και από πού προέρχονται. Έχω να σας κάνω λοιπόν μία πρόταση. Με τον Φίλιπ Μαϊστάκ και τον Εμμανουέλ Μακρόν είχαμε σχεδιάσει ένα σχέδιο που θα ενέπλεκε τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία όσον αφορά την ε, ε, αποταμίευση ενέργειας καθώς επίσης και τις επενδύσεις ε, και που θα αφορούσε 350 ε, ε, δις. Δηλαδή στην ουσία εμείς προτείναμε ε, από τη μία μεριά να υπάρχει η νομισματική δημιουργία η οποία να μην χρησιμοποιείται μονάχα και να μην οφείλει μονάχα τις τράπεζες αλλά τελικά να δημιουργεί και καλύτερη ενέργεια. Συμφωνείτε με κάτι, θα το στηρίζατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας. Βεβαίως αυτό είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα το οποίο αφορά και την σταθερότητα και την ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε ε, αυτά τα χρήματα αναφέρονται σε ένα πολύ ευρύτερο πακέτο. Και όλα αυτά βεβαίως ακόμα βρίσκονται υποσυζήτηση. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε πρόγραμμα θα είναι αξιόπιστο όσον αφορά τη σταθερότητα και την ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά θα αφορά την πραγματική οικονομία όπως είπατε και εσείς. Κατά αυτήν την έννοια βεβαίως ε, η πρόταση που κάνετε ε, όσον αφορά την ε, Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη. Στην Επιτροπή Μπαρόζο 1 υπήρχε, έγινε αναφορά στα λεγόμενα ομόλογα έργου. Βεβαίως ξέρουμε ότι θα πρέπει κανείς να δει τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε τελικά να παράγουμε αυτά τα 300 δις και για να είμαι ειλικρινής θα πρέπει να ε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία να είναι πιο δυναμική και η οποία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ε, ε, έτσι ώστε να μην ασχοληθούν μονάχα θα, πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές ε, να ε, βρουν λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ευρωπαϊκά ταμεία γενικά με επενδύσεις ε, που θα αφορούν προγράμματα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν ε, και τράπεζες αποταμιευτικές και ταμεία τα οποία αφορούν συντάξεις, ασφαλίσεις κτλ. έτσι ώστε να φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Εύκοβιτς. Ξέρουμε ότι εσείς πάντα αγωνιστήκατε για μια βιομηχανική πολιτική η οποία θα ελάμβανε ε, υπόψη το κόστος της ενέργειας καθώς επίσης και την κλιματική αλλαγή. Και βεβαίως ε, το σημαντικό ζήτημα είναι η διασύνδεση ανάμεσα στο, ε, στο πακέτο για το κλίμα του 2020 και την αποτελεσματικότητα από την άλλη για το 2030 είπαμε ότι θα πρέπει οι λύσεις από τεχνική και οικονομική άποψη να μπορούν να είναι σωστές ε, και να μπορούν να λειτουργήσουν για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ότι οι βιομηχανίες οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους καλά δεν θα πρέπει να χρειαστούν ε, να ε, υπομείνουν επιπλέον ε, ε, μέτρα τα οποία θα απεραίαν από ένα σύστημα εμπορίας ανταλλαγής εκπομπών και ένα σύστημα το οποίο θα ήταν δωρεάν και το οποίο θα τους δημιουργούσε πρόβλημα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός έτσι ώστε να αντισταθμιστεί το κόστος του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών. Επίσης η παραγωγή ξένη παραγωγή, παραγωγή, Κινέζοι ας πούμε, οι οποίοι ε, εξάγουν προς την Ευρώπη, πιστεύετε ότι θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο φόρο, κάποιο δασμό ψηλότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη για τις προσπάθειές του να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και για το γεγονός ότι έχει θεσπίσει στόχους για την ε, σημασία της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάσει στο 20% του ΑΕΠ, του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κέριο. Τώρα, όταν πρόκειται για το μέλλον της βιομηχανίας στην Ευρώπη, για την, ε, το ρόλο της ενέργειας στη βιομηχανία υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Το κόστος της ενέργειας και το κόστος του ηλεκτρισμού. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Αν δείτε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χοντρικής, οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες με τις τιμές των Ηνωμένων Πολιτών. Στο επίπεδο όμως λιανικής αγοράς ενέργειας, στο επίπεδο όπου πωλείται στις επιχειρήσεις μας, η ενέργεια είναι πολύ ψηλότερη, είναι δύο ή τρεις φορές υψηλότερο το κόστος της ενέργειας. Μια αντίστοιχη κατάσταση ισχύει για το φυσικό αέριο. Δεν είναι το κόστος λοιπόν παραγωγής της ενέργειας, είναι το κόστος μεταφοράς της ενέργειας, είναι η φορολογία της ενέργειας, και εμείς ουσιαστικά μειώνουμε την ανταγωνιστικότητά μας γιατί δεν έχουμε διασυνδέσεις, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστών για την ε, <clears throat> μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα άλλο σημείο που τόνισε ο κύριος Ταγιάννη είναι και αυτό πολύ εύστοχο και θα είναι και μία από τις κλίδες επιτυχίας εάν υπάρξει επιτυχία το, την Παρασκευή είναι το να εμποδίσουμε τη λεγόμενη διαρροή άνθρακο, δηλαδή τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σαφέ ότι ο μηχανισμός για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα θα πρέπει να παραμείνει στην εργαλειοθήκη μας, <clears throat> όχι για τώρα μονάχα, αλλά και για το διάστημα επέκεινο του 2020, αλλιώς οι επιχειρήσει μα θα μεταβούν σε άλλε χώρε όπου δεν υπάρχει σεβασμό. Ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα έχουν τη δυνατότητα να ρηπαίνουν περισσότερο και φυσικά με τον τρόπο αυτό χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας και τις θέσεις απασχόλησης. Ο κ. Εντουάρ να έχει το λόγο. Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά. Κύριε Σεφτσοβιτς, εδώ είμαι. Το χαρτοφυλάκιό σας έχει σαν τίτλο «Η Ενεργειακή Ένωση». Όπως ξέρετε και φάνηκε και με την ακρόαση της κυρίας Μπράτουσεκ, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το περιεχόμενο μιας τέτοιας ένωσης. Πέραν της συνθηματολογίας, τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η Ένωση και πώς θα μας βγάλει από την τωρινή κατάσταση, γιατί αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα συνδυάσετε την εθνική, πώς θα συμβάσετε μάλλον την εθνική κυριαρχικότητα στην πολιτική ενέργεια και την αυξανόμενη σύγκληση που είναι απαραίτητη για να υπάρξει μια κοινότηση, μια ένωση στον τομέα της ενέργειας. Λέτε ότι θέλετε να έχετε ένα τρίτο πακέτο. Έτσι θα το κάνετε αυτό ή θα περιμένετε να υπάρξει ενσωμάτωση και ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας από τις ίδιες τις αγορές. Και πώς θα μπορέσετε να επηρεάσετε την πολιτική των κρατών μελών με ένα είδος ε, ευρωπαϊκού εξαμήνου ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Σεύτσοβιτς, για το ερώτημά σας. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η τελική μορφή της Ενεργειακής Ένωσης από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μια συζήτηση σε βάθος και μαζί σας και με τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για την σωστή επεξεργασία μια πρόταση για την Ενεργειακή Ένωση και θα επανέλθω ενώπιον τη Επιτροπή σα για να το παρουσιάσω σε πιο λεπτομεριακό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι το τωρινό status quo είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να βελτιώσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν για μια μεγαλύτερη ασφάλεια στο ενεργειακό επίπεδο και για να αναπτύξουμε καλύτερα ένα μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα της οδηγίας για την ασφάλεια τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο. Πρέπει να διερευνήσουμε και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε επέκεινα του τρίτου πακέτου και πέραν των τωρινών ρυθμίσεων που ισχύουν. Γιατί θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ του υλικού και του λογισμικού ούτως υπήν σε ό,τι αφορά την υποδομή ενέργειας στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε καλή αποθήκευση φυσικού αερίου, καλή διασύνδεση, αυτό είναι το υλικό αν θέλετε, καλά λειτουργούντα και ευφυή δίκτυα στην Ευρώπη, αλλά και το λογισμικό τη ενέργεια είναι σημαντικό. Πολλέ φορέ βλέπουμε ότι επειδή δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, διαχειριστών των δικτύων και επειδή έχουμε διαφορετικούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο, διαφορετική μεθοδολογία, είναι πολύ περιορισμένο το εμπόριο ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση σε προσεγγίσεις. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να εξασφαλίσουμε ότι οι διαχειριστές των συστημάτων μετάδοσης ηλεκτρισμού και οι ρυθμιστές είναι πράγματι ανεξάρτητοι και έχουν τα κίνητρα να συνεργαστούν μεταξύ τους γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα πραγματικά ωφέλη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δική μου γλώσσα. Γιατί φυσικά και αυτή είναι μια γλώσσα που βρίσκεται στις δικές σας γλωσσικές δεξιότητες. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ ήμουν παρόν και στην ακρόαση στην Επιτροπή Μεταφορών όπου ήσασταν και εσείς παρόν την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν λαμπρή η παρουσίασή σας εκεί. Πιστεύω ότι και για τον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ενεργητικότητα και την ορμή που δείξατε σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τώρα, βέβαια, η συνδίκη τη Λισαβόνα λέει ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα να αποφασίσουν σε σχέση με το μείγμα ενέργεια που χρησιμοποιούν. Πώ θα μπορέσετε λοιπόν να συνδυάσετε και να συμβιβάσετε τα συμφέροντα των μεμονωμένων κρατών μελών ώστε να αποφύγουμε ένα κράτο μέλο να υφίσταται πιέσει ή να επηρεάζεται αρνητικά από τα άλλα κράτη-μέλη από την Κομισιόν. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικέ γεωγραφικέ συνθήκες, διαφορετικά, διαφορετικές ιστορικές παραδόσεις και όλα από αυτό μπορεί να αποκύψει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σεφτσοβιτς στα Σλοβακικά. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τη, στην πολιτική μεταφορών, Σας ευχαριστώ. Έχω τώρα μία νέα ε, θέση για την οποία είμαι υποψήφιος ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τα ενεργειακά θέματα. Αλλά φυσικά υπάρχει στενή σύνδεση αυτής της πολιτικής με την πολιτική μεταφορών. Θα πρέπει να τύχουν κοινού συντονισμού αυτές οι πολιτικές οι μεταφορές και το διάστημα φυσικά θα πρέπει να συνδυάζονται και να συντονίζονται με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρισκόμαστε σε ένα κοινό πλαίσιο και έτσι να τα, τις αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το δεύτερο σας τώρα ερώτημα, για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Είναι αλήθεια ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να επιμένουν ότι θα πρέπει να τηρηθεί η συνδίκη της Αβώνας σε ό,τι αφορά το δικαίωμά τους να προσδιορίσουν το περιεχόμενο της ενεργειακής τους πολιτικής και να παραμείνουν ανεξάρτητα και κυρίαρχα για τον προσδιορισμό του ενεργειακού μείγματος. Αλλά το ενεργειακό αυτό μείγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως θέμα συζήτησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι βέβαια βάσει τη συνθήκη στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, στην αποκλειστική αρμοδιότητα το θέμα τη ενέργεια για τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε ήδη μια εσωτερική αγορά και έχουμε καταφέρει να περάσουμε τρία πακέτα για τα ενεργειακά θέματα. Ω εκ τούτου, στον τομέα τη ενέργεια νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία και πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία ώστε να εξασφαλίσουμε λοιπόν τις διασυνδέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό συμφωνίες πλαίσιο, πλαισιού. Χέλβεκ Πέτερσον. Ναι, ε, θα είμαι... Ε, ε είμαι... Not only web it's also a 360 degree hearing. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, χάρηκα που είπατε ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ε, ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αντιμετώπισης κλιματικής ε, μεταβολής και της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, ε, είπατε ότι θα ενδιαφέρεστε τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο για το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής. Επίσης, ε, αναφερθήκατε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θεωρώ και εγώ ότι είναι το κλειδί για τη λύση του προβλήματος. Είπατε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα θα πρέπει να εξεταστεί ως πρώτη πηγή ενέργειας. Το ερώτημά μου είναι πώς θα πείσετε τις χώρες μέλη ότι πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο γιατί δεν φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την άποψη αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ πείτε μας κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Ε, πιστεύω πράγματι ότι το επιχείρημα εδώ είναι πολύ απλό. Ε, μπορούμε να δαπανίσουμε το 46% της ε, ενέργειας, ε, του λογαριασμού της ενέργειας για την θέρμανση και την ψήξη των κτηρίων μας δεν είναι υπερβολικά δαπανηρό όταν πληρώνουμε 400 δις ευρώ το χρόνο για την ενέργεια ε, πώς μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε την αποδοτικότητα στα κτίρια μας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Όταν ε, μελέτησα τις πολιτικές αυτές και επίσης ε, ρώτησα τους συναδέλφους και τους εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή γιατί είναι τόσο δύσκολο να πείσουμε τις χώρες μέλη και δεν μπορούμε να σημειώσουμε καμία πρόοδο ε, γιατί κατά μέρη η επιλογή είναι πολύ προφανής, εξόθαλμη. Μια από τις απαντήσεις ε, που νομίζω ε, δείχνει προς σωστή κατεύθυνση είναι το ότι μέχρι τώρα είχαμε υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των, κτηρίων θεωρείται μια υποχρέωση και ήταν ένα περιοριστικό, ρυθμιστικό πλαίσιο αυτό το οποίο κυριαρχούσε εδώ. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε περισσότερο ε, στην κατεύθυνση της παροχής κινήτρων. Δηλαδή πολίτες που θέλουν να έχουν μια πιο αποτελεσματική θέρμανση, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης στα νοικοκυριά τους. Γιατί ε, έχουμε καλά μοντέλα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την παροχή κινήτρων προς τους Δήμους και τις κοινότητες για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων ούτω ώστε οι χώρες μέλη πραγματικά να πάρουν πιο σοβαρά αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σακοράφα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε, μια ακόμη επίπτωση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σας είναι η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας κοινωνική κατηγορία, αυτή των ευάλωτων καταναλωτών στον τομέα τη ενέργεια, οι οποίοι πλήττονται από μια νέα και πρωτόγνωρη μορφή φτώχεια την ενεργειακή φτώχεια. Γνωρίζετε την έννοια τη ενεργειακή φτώχεια. Αδυναμία στοιχειώδου πρόσβαση στι απαραίτητε μορφέ ενέργεια που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπέ επίπεδο ζωή. Και μιλώ για το αυτονόητο. Πρόσβαση στο φωτισμό, ...στη θέρμανση, στην ψήξη, δηλαδή στις ελάχιστες παροχές που θα έπρεπε να παρέχονται σε όλους αδιακρίτως, αλλά εσείς τις αντιμετωπίζετε σαν εμπορεύματα. Ερωτώ λοιπόν και θα σας παρακαλούσα για συγκεκριμένη απάντηση. Η περιβόητη ενεργειακή ένωση που φιλοδοξείται να επιτύχετε με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου. Έχει τελικά χώρο για αυτή την κοινωνική τάξη ενεργειακής φτώχειας. Και αν ναι, πώς σκοπεύετε να κάνετε πράξη την κοινωνική, την αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, με ποιον ακριβώς τρόπο, ποια χρηματοδοτικά εργαλεία, τι ύψος πόρων και πόσο άμεσα σκοπεύετε να υιοθετήσετε και να τα διαθέσετε για να προστατεύσετε τους ευάλωτους καταναλωτές από την άνοδο των τιμών και τη συρρήκνωση των εισοδημάτων τους που τους οδηγεί στην ενεργειακή φτωχοποίηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου για αυτή την ερώτηση γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει χειροτερέψει το ζήτημα αυτό λόγω της ε, κρίσης και υπάρχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που είναι στερημένοι από την, ε, ε, που δεν και το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αν σκεφτούμε τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου θα πρέπει να πούμε ότι λόγω ακριβώς της πρόσφατης ε, κρίσης υπάρχει και περισσότερη ενεργειακή φτώχεια και στην Ευρώπη. Ε, μας ρωτάτε τι, τι, θέλουμε να κάνουμε. Ε, ξέρετε ότι όταν το θέμα είναι κοινωνική πολιτική, αυτό, η κοινωνική πολιτική είναι πάρα πολύ στις χώρες μέλη. Ε, από, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως ε, μπορούμε να διδαχθούμε ημένα από τους δε ε, όσον αφορά τη χάραξη μιας κοινωνικής πολιτικής για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τους πιο ευάλωτους πολίτες. Υπάρχουν διάφορα ε, μοντέλα στις χώρες μέλη και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε ποιο είναι το πιο ενδεδειγμένο μοντέλο για ποια χώρα. Ε, σε ορισμένε περιπτώσει άμεσα είναι σχέσει για τι ευάλωτε ομάδε ε, πληθυσμού. Ε, σε άλλε περιπτώσει οικονομική υποστήριξη για αυτού που δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό. Σε άλλες χώρες υπάρχουν κατόφλια όσον αφορά τις βασικές ανάγκες ενέργειας για τις πιο ευάλωτες ομάδες και πάλι του πληθυσμού. Όλα αυτά είναι μοντέλα που θα μπορούσαμε να αναλύσουμε συνεργασία με τις χώρες μέλη θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα, το κοινωνικό ταμείο, τα διαρθρωτικά ταμεία κλπ. Και είναι σημαντικό επίσης να υπάρξουν ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις γιατί θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη και οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές. Ε, κυρία Έγκστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφια πρόεδρε Σεύκοβιτς. Ε, θα ασχοληθώ με το ίδιο θέμα. Οι κλιματικοί στόχοι είναι πολύ καλή. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και να μειώσουμε ε, το ε, κάρβουνο. Αλλά σε μερικές χώρες ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επένδυση σε ανανεώσιμες. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ακούσαμε ότι τα ορυκτά καύσιμα θα έχουν περισσότερες επιδοτήσεις από, τα, από τις ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει όλο και περισσότερο και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ε, τα μέτρα για την ανάπτυξη των ε, εναλλακτικών μορφών ενέργειας θα αντιμετωπίσουν και την ενεργειακή φτώχεια. Ε, δύσκολο το ζήτημα και όχι απλή απάντηση. Αυτά είναι σημαντικές προκλήσεις και για τα κρατη και για την Κομισιόν αλλά και για την Ένωση. Ε, όσον αφορά το μέλλον. Το πρώτο σκέλος της απάντησής μου θα είναι το εξής, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά ενέργειας, ε, γιατί εάν δει κανείς ε, τις τιμές χονδρικής για την ενέργεια, είναι συγκρίσιμες με αυτές ε, που βλέπουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μερικές φορές όμως βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ε, ηλεκτρισμού στις αγορές μας αλλά ε, δεν υπάρχουν αρκετές κοινέ προσπάθειες, δεν υπάρχουν TSOs, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει συντονισμός και ρύθμιση και επομένως μονάχα με την ενιαία αγορά θα καταφέρουμε να έχουμε όλα αυτά τα ωφελήματα τα οποία θα μειώσουν προς τα κάτω, θα πιέσουν συγγνώμη προς τα κάτω τις ε, ε, τιμές ε, της, του ηλεκτρικού. Η δημόσια παρέμβαση στον τομέα της ενέργειας είναι 120-140 δις το χρόνο. Είναι πολλά χρήματα Δηλαδή γίνονται και υπάρχουν τα συστήματα ε, επιδότησης αλλά παρόλα αυτά παραπονιέται ο κόσμος. Το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει από τη μία να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι περιορισμοί της ε, ενιαίας αγοράς ενέργειας θα αρθούν έτσι ώστε να ωφεληθούμε πραγματικά από αυτή την νέα αγορά ενέργειας. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ έντιμη συζήτηση όσον αφορά την δομή ε, της ενέργειας ε, ε, και της αγοράς ενέργειας και να είμαστε πάρα πολύ στην Ευρώπη και να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όσον αφορά τις δυσκολίες οι οποίες ακριβένουν πολύ και την ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ Ζόρταν Μπαλόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεύτσοβιτς. Έχετε πίσω σας μια εντυπωσιακή πορεία και έχετε μια μεγάλη εμπειρία για τα εξωτερικά θέματα ως διπλωμάτης. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, η κυρία Βιελίτσοκο και αυτή έχει ε, βρεθεί εκεί. Έχετε περάσει κι εσείς και έχετε μια μεγάλη εμπειρία για τη διαχείριση, για θέματα διαχείρισης σε υψηλό επίπεδο. Εσείς αν σας έλεγε κάποιος να γίνετε καπετάνιος σε ένα υπεροκιάνιο, θα το κάνατε αυτό με την εμπειρία σας. Και τώρα είσαστε έτοιμος εσείς να διευθύνετε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε μεγάλο ταλέντο, μπορείτε να ετοιμαστείτε σωστά για τις ακροάσεις, να απαντήσετε τα ερωτήματα αυτά. Αλλά αν αναρωτιέμαι, είναι τόσο πολύπλοκο ο τομέα της ενέργεια. Μήπως θα έπρεπε να έχετε ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε αυτό το θέμα, δεν θα ήταν πιο τολμηρό από εσά να το αναγνωρίσετε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Σεφτσεβιτ. Αναγνωρίζω ότι η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κέρια. <clears throat> Και πιστεύω ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη μας έχουν μια μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στα θέματα αυτά. Αυτό το οποίο χρειάζεται στον σημαντικό τομέα αυτό και στην, στον ευραλικό αυτό τομέα χρειαζόμαστε πολιτική θέληση, χρειαζόμαστε ηγετικό ρόλο, χρειαζόμαστε τις διπλωματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη μας να ξεπεράσουν την ε, περιχαρακωμένη τους κυριαρχικότητα και να προχωρήσουν σε μια ενεργειακή ε, ένωση και χρειάζεται κανείς να έχει την ικανότητα να διαπραγματεύεται με τους τόσο σημαντικούς αυτούς εταίρους και αντιπάλους όπως είναι η Ρωσία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χρειάζεται λοιπόν να έχει κανείς εμπειρία εξωτερικών σχέσεων για τις διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους για την ε, σφυριλάτηση μιας πολιτικής εναντί της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύετε ότι θα είχε ότι υπάρχει ένας χώρος όπου υπάρχουν περισσότερα διακυβευόμενα από ότι η συνδιάσκεψη του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή. Πιστεύω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση δεν δεν απόκειται μόνο σε μένα και στον Επίτροπο για την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι θέμα και για την κυρία Μογκερίνη ως εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο προτεραιότητας για την ενεργειακή διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είμαι λοιπόν απόλυτα έντιμος απέναντί σας, πιστεύω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δική μου εμπειρία και τα τις γνώσεις μου σε επίπεδο εξωτερικών υποθέσεων με τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες. Είμαι σίγουρος θα με υποστηρίξουν οι υπηρεσίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη στο ρόλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, υποψήφια Αντιπρόεδρε για τις απαντήσεις σας. Ζητώ τώρα από τον συναδελφό μου, τον κύριο Λαβία, να προεδρεύσει του δευτέρου τμήματος της ακροασής μας. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε το σύστημα ping-pong με το ερώτημα της κυρίας Κιώστιγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε πει πολλά ήδη για τις ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά ίσως θα πρέπει να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Κομισιόν στην οποία εσείς ήδη συμμετέχετε και θα συμμετέχετε και στο μέλλον, έχει ε, υποστηρίξει τις επιδοτήσεις για το Hinkley Point, ένα σταθμό πυρηνικής ενέργειας στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζετε ότι είναι σαφής οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η δημιουργία ε, ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να είναι το προέχον στα, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Για μας είναι σαφές ότι εδώ βλέπετε να είμαστε ενώπιον μιας ε, επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια σημαντική, μια τεράστια στρέβλωση ανταγωνισμού έναντι της ποινική ενέργειας έναντι των ανανεωσίμων ενεργειών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς θα, πώς, ε, τι θέση είχατε εσείς για την απόφαση της Κομισιόν για την έγκριση αυτών των επιδοτήσεων προς το Hinkley Point. Ευχαριστώ την απάντηση παρακαλώ κύριε υποψήφια επίτροπε. Σας ευχαριστώ κύριε Ακριστή για το ερώτημα αυτό και αυτό αξίζει πράγματι μία διευκρίνηση. Η απόφαση για το Hinkley Point δεν αφορούσε την προτίμηση στην πυρηνική ενέργεια εναντί ανανεώσιμη ενέργεια. Ήταν μια καθαρή περίπτωση κρατικής αρρωγή. Ήταν λοιπόν μια υπόθεση την οποία είχε αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Οι Βρετανικέ Αρχές παρουσίασαν ε, πιστικά επιχειρήματα για να μπορέσουν να δοθούν αυτές οι κρατικές επιδοτήσεις στο σταθμό του Hinkley Point έδωσαν σαφή στοιχεία βάσει των οποίων προκύπτει ότι θα θέλανε 7% της ε, ενέργειας να καλυφθούν από τον σταθμό του Χίγκλιπον, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα είχαν προβλήματα στην αγορά ενέργειας, δεν θα μπορέσουν να έχουν την απαραίτητη ε, χρηματοδότηση από τις χρηματαγορές για τη δημιουργία ενός σταθμού χωρίς την κρατική επιδότηση. Ήταν μια πολύπλοκη λοιπόν διαπραγμάτευση που έγινε με τις Βρετανικές Αρχές και η Κομισιόν επέμεινε στο να, υπάρχουν, να υπάρξουν οι καλύτεροι δυνατοί όροι για τους Βρετανούς καταναλωτές και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με το κόστος αυτού του εγχειρήματος οδήγησε σε χρηματοδότηση 70% από το κράτος, 30% από τους ιδιωτικούς επενδυτές με πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές από τις στις αρχές των ε, διαπραγματεύσεών μας όταν παρουσιάστηκε αυτό το θέμα στην ε, υπηρεσία ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Πανιό Κύριε αντι... Οψήφια Αντιπρόεδρε, εγώ βρισκόμαι εδώ, είμαι από την άλλη πλευρά. Καταρχήν θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ για την ενεργητικότητά σας, για την μεγάλη σας θεληματικότητα. Και στα εισαγωγικά σας λόγια είπε, είπατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την Ενεργειακή Ένωση, είπατε ότι θα έπρεπε να είχε διαμορφωθεί ήδη από πολύ καιρό, μιλήσατε και τους πέντε πυλώνες, ε, και ε, βεβαίως γνωρίζουμε ε, όσον αφορά τους στόχους αυτούς ε, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης αυτών των στόχων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είστε υπέρ μιας ενεργειακής ένωσης όπως αυτή που προσεγγίζει ο κύριος Ντόναλτ τους Τάσκ, ο νέος ε, πρόεδρος του Συμβουλίου ή πρόκειται για μια κοινή αγορά φυσικού αερίου έτσι όπως την πρότεινε ο Ζακ Ντελόρ αλλά και ο κύριος ε, Μπούζεκ εμπνεόμενος από την ε, Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να κατάλαβα καλά την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει διαφορετικά, διαφορετικές αφετηρίες που οδήγησαν στην ε, συζήτηση αυτή, στο διάλογο αυτό. Πιστεύω ότι η Ενεργειακή Ένωση ήταν ε, ένα μοντέλο ε, των φιλοευρωπαϊστών όπως ο Γέρζι Μπούζεκ και ο Ζακ Ντελόρ, στους οποίους αναφέρθηκα άλλωστε και υπέρξαν και άλλοι πολιτικοί οι οποίοι ε, είχαν προτείνει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και μια από τις πιο πρόσφατες προτάσεις προέλθε από τον μελλοντικό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Ντόναλτ Τούσκ για να το προφέρω σωστά. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα συμβεί στο τέλος είναι το εξή. Θα παρουσιάσω το δικό μου πολιτικό μοντέλο που θα βασίζεται σε αυτούς τους πέντε πυλώνε. Ενδεχομένω αν τέσσερι θα τροποποιηθεί, αλλά θα ήθελα να έχουμε έναν διάλογο να σχέση με το πώ μπορούμε να πετύχουμε μια συνένεση όσον αφορά την δομή, τι πολιτικέ το ε, πλάνο δράσης, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματά μας σε, τακτικές, ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα ήθελα να σας πω όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου. Όταν διατυπώνει κανείς αυτή την πρόταση, αυτό το οποίο ακούει από τους αμπειρογνώμονες είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Υπάρχουν πολύ σύνθετες ε, κανόνες περί ανταγωνισμού, ε, σύνθετοι κανόνες του ΠΟΕ. Υπάρχουν κάποιες ε, ανησυχίες ε, σε θα έχουμε μια ε, διευθέτηση που θα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε περίπτωση χωριστά. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις αρχές ανησυχίες γιατί πιστεύω ότι το επιχείρημα του πόσο δαπανάμε σε ενέργειες, πόσο μεγάλος πελάτης είμαστε ε, μετράει και πραγματικά αξίζουμε καλύτερη μεταχείριση, καλύτερες τιμές και μεγαλύτερο σεβασμό Και τώρα η ερώτηση του κυρίου Τεμές Μέκερ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σεύκοβιτς. Εδώ είμαι. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είπατε ε, τώρα μόλις ότι είστε η υπέρ δεσμευτικών στόχων της ενεργειακής αποδοτικότητας και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω 100% μαζί σας. Ωστόσο είμαι κάπως απογοητευμένος ακούγοντας ε, τα αποτελέσματα της Ενάντησης κορυφής. Ε, δηλαδή οι επικεφαλής των κυβερνήσεων τελικά μίλησαν όχι για δεσμευτικούς αλλά για ενδεικτικούς στόχους. Ε, νομίζω λοιπόν ότι χάσαμε την ευκαιρία. Θεωρείτε ότι τέτοιοι ενδεικτικοί στόχοι τελικά θα έχουν τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Δεύτερον, η υποστήριξη ε, των ε, επιχειρήσεων ε, θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω. Πώς μπορείτε να το συνδυάσετε με τις πρωτογενείς επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη στήριξη των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Ε, βλέπω ότι έχετε μελετήσει πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα από τη συνάντηση κορυφής του Συμβουλίου και είναι αλήθεια ότι το σχέδιο των ε, απορισμάτων λέει, αναφέρει ότι όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα μιλάμε για ενδεκτικούς στόχους. Όπως σας είπα, αύριο θα ασκήσω πίεση ούτε ώστε οι στόχοι αυτοί να αποκτήσουν ένα δεσμευτικό χαρακτήρα. Αλλά ξέρετε ότι οι αποφάσει λαμβάνουν το Συμβούλιο μέσω συνένεση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ποια θα είναι η τελική έκβαση. Ωστόσο, θα ήθελα να σα πω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Δηλαδή, βασιζόμενο στην εμπειρία που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, την θέσπιση αυτών των στόχων και την ε, χάραξη πολιτικών στο τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Ε, καμία φορά είναι σημαντικότερα από τους στόχους τα συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές. Επίσης τα μοντέλα παροχής κινήτρων. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε στα χέρια μας, στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, ε, ε, το πώς εμείς θα επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα του Συμβουλίου και πώς θα τα μεταφράσουμε, θα τα μεταφέρουμε σε, συγκεκριμένες συγκεκριμένε πολιτικές. Νομίζω ότι είναι μια βασική προτεραιότητα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής η προβολή του επιχειρήματος του τεράστιου κόστους και των ενεργειακών απολειών ε, που έχουμε, καθώς και το εξαιρετικά υψηλό κόστος που πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες, για παράδειγμα, επειδή το κτίριο στο οποίο κατοικούν δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, στις γραπτές σας απαντήσεις είπατε, ε, αναφέρατε ε, την ε, πρόθεση άλλων μορφών πλήν των ορυκτών καυσίμων. Ίσως θα ξέρετε και από την Πρατισλάβα ότι δεν αποφασίζεται τόσο εύκολα και απλά αυτό. Αγγίζει κάποια πράγματα η Κομισιόν αλλά δεν τα προωθεί σε βάθος ερώτηση. θα βάλετε σαφείς στόχους ή θα αγγίξετε κάποια θέματα εσείς και κάποιοι άλλοι. Ε, νομίζω ότι αναφερθήκατε ε, ε, ε, εν τέλει στα βιοκαύσιμα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. ναι, κοιτάξτε. Εάν πάρω την έγκρισή σας ε, αυτό το ζήτημα οπωσδήποτε ε, θα μπει στο τραπέζι του διαλόγου. Ε, εάν προσέξει κανείς και την οδηγία σχετικά με την ε, χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης γης ε, θα καταλάβει ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και από το Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη αλλά ότι όλοι προσπαθούν να βρουν κάποιο κοινό τόπο όσον αφορά το θέμα αυτό. Είπατε αγγίζουμε πράγματα και δεν τα κάνουμε σε βάθος. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτή η γενιά των βιολογικών τροφίμων ε, και των βιολογικών ε, παραγωγών ε, που θα πρέπει να αντικατασταθούν από καλλιέργειες για βιοκαύσιμο δεν έχουν μελετηθεί ακόμα πολύ. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν επίσης και κάποιες κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες δεν είχαν αντιμετωπιστεί, δεν είχαν προβλεφθεί. Είναι γεγονός γεγονός ότι μπορούμε να κινητροδοτήσουμε τους ε, ερευνητές έτσι ώστε να μελετήσουν περισσότερο την δεύτερη ε, γενιά των ε, βιοκαυσίμων γιατί όντως θα τα χρειαστούμε στο μέλλον αλλά μπορούμε, μπορώ επίσης να σας πω ότι πιστεύω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα δούμε κυρίως ε, στον τομέα των μεταφορών ε, ευρύτερη χρήση εναλλακτικών ε, μορφών ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια κτλ. έτσι ώστε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε και στα βιοκαύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Γερίστια Μπαούνσε. Καλησπέρα κύριε Σεύκοβιτς, Σεύκοβιτς, στα αριστερά σας, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, θα ήθελα για το σταθμό της ε, Χαρόνια, ο οποίος είναι από τους παλιότερους της Ισπανίας και βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, στην ε, ε, Βιτόρα Γκαστέιτς ή στο Μπιλμπάου και η οποία έχει θεωρηθεί ότι είναι ε, επικίνδυνοι όπως κάποιοι άλλοι σταθμοί που έτρεψαν στο Βέλιο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό, η Ισπανική κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτό το σταθμό. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά η ασφάλεια των ενεργειακών σταθμών είναι δικό σας, προ, σας θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν εσείς είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το θέμα των πεπαλαιωμένων πυρηνικών σταθμών ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι το θέμα της ασφάλειας ε, το, των πυρηνικών εγκαταστάσεων το ζήτημα, ε, αυτό το ζήτημα είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε στενά με την Ισπανική κυβέρνηση στην Κομισιόν έχουμε 180 ενεργεια πυρηνικούς ε, επιθεωρητές έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια και με υψηλά πρότυπα. Τα stress tests τα οποία κάναμε μετά την ε, τραγωδία της Φουκουσίμα έδειξαν πρόσφατα αλλά και βέβαια όλη η πραγματογνωμοσύνη που έχουμε στην Κομισιόν ότι μας απασχολεί η ασφάλεια και ε, ότι ε, διασφαλίζεται αυτή η ασφάλεια εάν υπάρχουν ή σε περίπτωση που υπάρξουν οποιασδήποτε αμφιβολίες από πλευρά της Κομισιόν όσον αφορά την ασφάλεια ή την ασφαλή λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων τότε οπωσδήποτε θα έρθουμε σε επαφή με την Ισπανική κυβέρνηση ε, και σε έναν ανοιχτό διάλογο αλλά με σαφή στόχο θα ε, πούμε στην ε, Ισπανική κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έριξον. Καλησπέρα κύριε Σεύκοβιτς. Από τη Σουηδία λοιπόν είμαι. Σουηδία 10 βαθμούς λέει ο μιλητής. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ένωση ενέργειας και ότι θα πρέπει να αναλυφθούν τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να το επιτύχουμε. Αλλά Ένωση Ενέργειας ε, θα πρέπει να, αυτή η ένωση θα πρέπει να βασιστεί στην ε, αλληλεγγύη και η κατάσταση είναι δύσκολη. Ας πούμε στη χώρα μου Έχουμε επενδύσει σε ε, θερμοηλεκτρικούς σταθμούς πριν από 100 χρόνια περίπου ε, και τώρα έχουμε τη δυνατότητα για ανανεώσιμες ε, πηγές και ε, επενδύουμε και επενδύουμε πολύ και για την ενεργική αποδοτικότητα και στην ε, βιομηχανία αλλά υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το κάρβουνο ας πούμε, τον άνθρακα. Ε, τι προτίθεστε να κάνετε. Απάντηση παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, έχετε δίκιο ότι η ελληνική και η εμπιστοσύνη, θα προσθέσω εγώ, είναι απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την ε, Ενεργειακή Ένωση της Ευρώπης. Ε, είναι πολλά και δύσκολα τα προβλήματα και υπάρχουν στιγμές όπως το 2009 όπου τα προβλήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα ε, επομένως εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε ε, να μπορέσουν ε, οι χώρες να έχουν την ενέργεια, το φωτισμό, τον ηλεκτρισμό που χρειάζονται. Η Σουηδία βεβαίως ε, είναι από τους πιο καλούς μαθητές. Πρέπει να συγχαρούμε την χώρα όσον αφορά την δομή της ε, ενέργειάς της και όσον αφορά την χρήση ανανεώσιμων ε, πηγών. Βεβαίως έχουν και τις γεωγραφικές συνθήκες που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές και το έκαναν με μεγάλη τεχνογνωσία και με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ε, σήμερα βεβαίως πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί και να πούμε ότι ο άνθρακας εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερο από το 27% της ενέργειάς μας παράγεται από άνθρακα. Μετά έρχεται η πυρηνική ενέργεια και πολύ πίσω οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επομένως έχετε δίκιο ότι περισσότερο από το 80% της ενέργειάς μας ε, δημιουργείται από το από τον άνθρακα, 44% ας πούμε της ενέργειας της Γερμανίας παράγεται από άνθρακα και λέτε τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, έναν, ε, μια νέα τεχνολογία όσον αφορά την ε, όσον αφορά τον άνθρακα όσον αφορά την συγκράτηση και την αποθήκευση του άνθρακα θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας για αυτά σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Βιρκούνεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Σεύτσοβιτς είπατε προηγουμένως το είπατε κατά επανάληψη ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις ενέργειας πρέπει να εξυγχρονιστούν και να επεκταθούν για να μπορούν οι ενεργειακοί πόροι να κινούνται ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις ενεργειακές νήσους μέσα εισαγωγικά. Αλλά έχουμε πολλές τέτοιες νησίδες και στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης από όπου προέρχομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θεωρείτε τα πιο κατεπήγοντα σχέδια, τα πέντε πιο κατεπήγοντα σχέδια για την ε, ενεργειακή ε, πολιτική της Ευρώπης και πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πέντε σχέδια κατά την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ γιατί αν δείτε την κατάσταση των ενεργειακών νήσων έχουμε σίγουρα ένα πρόβλημα στη, στο Βορρά, στην Φιλανδία, στα Βαλτικά κράτη όπου βλέπουμε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι συνδεδεμένα στις πηγές του παρελθόντος Έχουμε προβλήματα επίσης στην ε, νησιωτική ε, Ευρώπη, στη Μάλτα, στη Γύπρο, στα νησιά της Ιβηρικής Χεσονησό. Μου πείτε ποια είναι λοιπόν τα πέντε βασικά σχέδια για το μέλλον. Θα σας έργα, για μένα η καλύτερη απάντηση θα είναι να δείτε τον κατάλογο των σχεδίων τα οποία έχουν προσαρτηθεί στον ε, κατάλογο για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια και από εκεί θα δείτε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε διασυνδέσει μεταξύ Φιλανδίας και Βαλτικών χωρών και των υπολείπων χωρών της Ευρώπης για την διανομή ηλεκτρισμού. Αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη βδομάδα νομίζω θα ξεκινήσει ο ενεργειακός σταθμός της Κλαϊπέδας που είναι πολύ σημαντικός ως τμήμα αυτής της προσπάθειας να ξεπεραστεί αυτή η απομονωμένη ε, κατάσταση των Βαλτικών και ε, σκανδιναβικών κρατών, ενώ την ε, Φιλανδία περισσότερο. Θα έλεγα λοιπόν ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Φιλανδίας και Βαλτικών κρατών και επίσης ενεργειακή τερματική σταθμή στην περιοχή από όπου προέρχεστε και εσείς. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε έτσι να ξεπεράσουμε την ε, απομόνωση των περιοχών και θα βοηθήσει και τη Φιλανδία και τα Βαλτικά κράτη σιγά σιγά να ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενέργειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλλος Ζουρίνιου. Εδώ είμαι κύριε ε, υποψήφιε αντιπρόεδρε έχετε ένα πάρα πολύ σημαντικό καθήκον, μια σημαντική αποστολή, να μπορέσετε να βάλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο πρωτοπόρου για την πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες ενέργειες και συγχρόνως να εξασφαλίσετε την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα. Τρία ερωτήματα. Πρώτον, για το πακέτο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό το 27% για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Δεν θεωρείτε ότι το 30% θα είναι μεγαλύτερη αξιοπιστία στις δηλώσεις του Ζαν Claude ότι η Ευρώπη θέλει να είναι πρωτοπόρος και ηγέτης στις ανανεώσιμες ενέργειες. Δεύτερον για τις διασυνδέσεις έχουμε για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη πρέπει να έχουμε καλές διασυνδέσεις ενέργειας. Πώς θα μπορέσετε να το επιτύχετε αυτό, ιδίως στην περίπτωση της ε, Ιβηρικής Χερσονήσου, η σύνδεση με την Γαλλία Τρίτον, υπάρχουν ορισμένε κυβερνήσει οι οποίε έχουν περικόψει αντί να αυξήσουν τα κίνητρα για τη χρήση ε, ανανεώσιμε ενέργειε. Ποια είναι η άποψή σα για αυτέ τι πρακτικέ αυτών των κρατών Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το τέλο τη ε, ερώτησή σα. Το πρώτο τμήμα ουσιαστικά το έχω απαντήσει ήδη. Είναι σημαντικό ότι η Πορτογαλία και η Ισπανία βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση γιατί δεν έχουν πετύχει ακόμα, είναι πολύ μακριά από το στόχο διασύνδεσης ενέργειας μεταξύ των μελών. Θα θέλαμε να είναι 10% αλλά μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας είναι μόνο 2 με 4%. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό, είναι απαράδεκτη κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε καλές απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα. Ήδη θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις την Πέμπτη και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα πρόβλημα προς λύση, ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σωστή χρηματοδότηση και τόσο η Ισπανία όσο και η Πορτογαλία θα πρέπει να μπορέσουν να συνδεθούν πλήρω με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Η Κομισιόν, όπω σα είπα, είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή, όχι μόνο για αυτό το πρόβλημα, αλλά και για άλλε περιπτώσει όπου βλέπουμε ότι σε περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ να μπορέσει να εξευρεθεί μια Είμαι έτοιμο λοιπόν να συμμετάσχω στι διαπραγματεύσει αυτού του είδου γιατί νομίζω ότι αυτέ οι καταστάσει θα πρέπει να ξεπεραστούν. Δεύτερο πρόβλημα που θέτεται είναι και αυτό σημαντικό. Έχουμε μια κατάσταση στην Ισπανία, την Πορτογαλία, επίση και στη Τσεχική Δημοκρατία όπου έχουν εγκριθεί κάποια συστήματα για οικονομική υποστήριξη της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας. Και μετά αυτές οι πολιτικές έχουν αναστραφεί. Η Πορτογαλία για μένα είναι καλύτερο παράδειγμα γιατί εκεί έγινε μια διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων <clears throat> για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και υπήρξαν κάποιες συμβαστικές λύσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όμως τα πράγματα έχουν εμπλακεί σε πολύπλοκες νομικές μάχες σε σχέση με την ε, με τον αναδρομικό χαρακτήρα ορισμένων αποφάσεων. Εγώ θα προτιμούσα αντί να υπάρχουν νομικές διαμάχες να γίνουν πραγματικές διαπραγματεύσεις. Κύριε Βυσνιεύσικα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι το εξή. Ποια είναι η δική σας ε, θέση όσον αφορά στην ε, ε, διασύνδεση μεταξύ ενεργειακού πακέτου και ανταγωνιστικότητας ε, ε, και εξάρτηση, συγγνώμη. υπάρχει μεγάλη εξάρτηση Ευρώπης από τη Ρωσία. Η Πολωνία από την οποία εγώ προέρχομαι είναι και αυτή σε δινή θέση. εισάγουμε δύο ε, τα δύο τρίτα του αερίου. Αλλά ωστόσο η δική μας, και η δική μας ενεργειακή παραγωγή βασίζεται στον άνθρακα. Ε, θεωρείτε ότι έχει έρθει κατάλληλη ε, στιγμή για την χάραξη μιας ενεργειακή ε, πολιτική στην Ευρώπη που δεν αποκλεί ε, τις ε, πηγές του άνθρακα γιατί η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό ε, ε, από χαμηλό, χαμηλού κόστους άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η αντίφαση στη νέα ατζέντα ε, με τους στόχους ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τον ε, άνθρακα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα δύο να αναπτυχθούν παράλληλα και να ενισχυθούν αμοιβαία. Γιατί ε, όταν, όσον αφορά τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτές είναι ε, ε πηγές ενέργειας. Η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια. Ε, με τον τρόπο αυτό γινόμαστε πιο ανεξάρτητοι από την εισαγωγή ενέργειας, εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία κυρίως με την οποία σε αυτή τη συγκυρία βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε ε, και για τις δύο πολιτικές ταυτόχρονα και μπορούμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Όπως σας είπα, η απόφαση για το ενεργειακό μείγμα είναι μια κυρίαρχη απόφαση των χωρών μελών, αλλά ταυτόχρονα κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να σέβεται τους κοινού στόχους στους οποίους έχουν αποδεχθεί οι χώρες μέλη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή ε, για ε, την, τις πράσινες πολιτικές και για μια πιο πράσινη στρατηγική για το μέλλον. Ε, νομίζω ότι το πακέτο 2030 θα είναι θετικό για την Πολωνία γιατί υπάρχουν δύο σημαντικά πολιτικά στοιχεία σε αυτό το πακέτο. Πρώτον, η δημιουργία Ε, η ενίσχυση μάλλον της ε, έρευνας, και ε, έρευνας για, την, για μεθόδους δέσμευσης και αποθήκευσης της ενέργειας. Επίσης σταθμή συμπαραγωγής ενέργειας ούτως ώστε και η Πολωνία να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους στόχους στην ε, πράσινη ε, ατζέντα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, σε συνέχεια των απαντήσεων σας μέχρι στιγμής θα ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε ότι αναπόκειται στις χώρες μέλη να λάβουν τις αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Η ερώτησή μου έχει ως εξής πώς ε, σχεδιάζεται να... πώς προγραμματίζεται τη συνεργασία μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις ενεργειακές πολιτικές. Και θα ήθελα να μας πείτε κάτι πια πράγματα για την ε, δυνατότητα διαφοροποίησης ε, των πηγών παροχής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι, απάντηση, πιστεύω ότι ο καλύτερος συντονισμός και η διαφοροποίηση είναι παράγοντες κλειδιά στην ε, δημιουργία μιας ε, ενεργειακής ένωσης στην Ευρώπη. Χωρίς καλό συντονισμό και χωρίς ε, μια διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας δεν νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Όσον αφορά το συντονισμό νομίζω ότι έχουμε ήδη μια θετική εμπειρία με τις ομάδες συντονισμού για το φυσικό αέριο και νομίζω ότι εδώ έχει, υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνη ε, και υπάρχει όλο και περισσότερη διαφάνεια στις συναντήσεις της ομάδας. Και ε, νομίζω βεβαίως ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να είναι έντιμες όσον αφορά τις ε, συνθήκες διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή γραμμή στις επαφές με τις τρίτες χώρες για να εξασφαλίσουμε οι εταίροι μας να μην παίξουν στο χαρτί του διέρη και βασίλευε απέναντι στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο αυτό που ισχύει για την ε, ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο και για τις άλλες πηγέ ενέργειες. Τώρα, όσον αφορά τη διαφοροποίηση, το πρώτο στοιχείο κλειδί για το αέριο, ε, και έμαθα κάποια πράγματα από την αποτυχία του Ναμπούκο, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο, να έχουμε πια πιο συγκεκριμένη πολιτική παρουσία σε όλες τις χώρες εκεί όπου φτιάχνεται αυτός ο αγωγός του νοτίου διαδρόμου. Ε, επίσης θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επαφή με την εταιρεία η οποία φτιάχνει αυτόν τον αγωγό ε, και θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ε, υποστήριξη για τα έργα αυτά. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά τερματικά, τις νέες σχέσεις με την Αλγερία ή χώρες όπως είναι η Βραζιλία ή άλλες χώρες από τις οποίες επίσης θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε ενέργεια εφόσον βεβαίως ε, δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Σεύκοβιτσε, ε, χαίρομαι, χαίρομαι που μιλάτε ε, για αυτά τα θέματα. Υπενθυμίσατε και τις τους διαχωρισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και ότι βεβαίως η ενέργεια δεν πρέπει πια να χρησιμοποιείται σαν πολιτικό όπλο. Μιλήσατε και για τη Ρωσία. Θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα όσον αφορά την ενέργεια. Πώς θα διαχειριστείτε πώς προτίθεστε να διαχειριστείτε τις σχέσεις με την Ρωσία, κυρίως όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρετε ότι επί σειρά ετών η Ρωσία ήταν στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η κατάσταση στην Ρωσία είναι βεβαίως πολύ στρατηγική, αλλά οι εταίροι έχουν ε, διαφορετικές θέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς, ανοιχτοί και διάφανοι στις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Και θα πρέπει σαφώς να δηλώσουμε τη θέση μας όσον αφορά την, ε, τις ε, ε, ρωσικές εταιρείες οι οποίες επιχειρούν ε, στο ενωσί, στην ενωσιακή επικράτεια θα πρέπει σαφώς να σεβαστούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι Όσον αφορά, λέω, τον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ε, ε, δυνατότητα που έχει η Ευρώπη ή που πρέπει να έχει για μια συνολική αγορά. 52% ε, του, των εσόδων της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφορά την, τα προϊόντα ε, ενέργεια. Δεν είναι δηλαδή ότι από την καλή τους καρδιά εξάγουν ενέργεια σε εμά. Ε, είναι απαραίτητη αυτή η εξαγωγή για τη χώρα. Θα πρέπει να διευρύνουμε λοιπόν τη σχέση και θα πρέπει σαφώς να μπορούμε να μιλάμε με μία φωνή όπως συνέβη φέτος. Ο πρόεδρος Πούτιν έστειλε ας πούμε 18 επιστολές σε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ο κύριος Σεβδάνης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ οι απαντήσεις σας είναι πολύ ενθαρρυντικές ε, και χαίρομαι που θα συμμετάσχετε ε, στο, στη διάρκεια του Παρισιού και βεβαίως ε, πολύ ενθαρρυντικές είναι και οι γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε. πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να έχετε πλήρη ρόλο στο Παρίσι. Σε σχέση με την κλιματική πολιτική, τι θα κάνετε έτσι ώστε ε, να μην ασχοληθεί μόνο με το κλίμα η συζήτηση στο Παρίσι και τι θα κάνετε έτσι ώστε ε, να ε, συνεχίσουν σωστά οι διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια των ΗΠΑ και να καταλήξουν σε δεσμευτικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σας απαντώ αμέσως όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την διάσκεψη του Παρισιού και την ίδια τη διάσκεψη. Όπως και σε προηγούμενες διασκέψεις βεβαίως, ξέρουμε ότι η εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ε, μεγάλη, θα είναι επίσης ε, πολύ προσεκτική ε, όσον αφορά τις συζητήσεις και βεβαίως και όσον αφορά και το και βάση και του ε, της συμφωνίας πλαισίου που διαπραγματεύονται το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν είναι σαφής, είναι ο μηχανισμός, είναι καθαρός για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πληροφορείται την ε, ε, έκβαση των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως θα διασφαλίσω τη σωστή σας διαβούλευση και πληροφόρηση στον δρόμο προς ε, το, τη διάσκεψη κορυφής ε, του Παρισιού. Όσον αφορά τώρα την ενίσχυση της ε, στήριξης των πράσινων πολιτικών και των ανανεώσιμων των πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το ζήτημα και τα κράτη-μέλη οπωσδήποτε, ότι το ζήτημα δεν αφορά μονάχα την προστασία του περιβάλλοντος, είναι και οικονομικό ζήτημα. Μας δίνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μας βοηθάει όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, ε, δημιουργεί θέσεις εργασίας γιατί ε, ήταν πραγματικά ε, ένας από τους λίγους τομείς που κατάφερε να κρατήσει τις θέσεις εργασίας. Επίσης ξέρουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία, τεχνικές ε, γνώσεις καλές και είναι γεγονός ότι σε, χώρες, σε σχέση με χώρες όπως η Κίνα ας πούμε είναι γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αναπτύξει σημαντική τεχνολογία, πράσινη τεχνολογία. Ευχαριστώ. Μαρι... Ζαν Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε για τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά σίγουρα για τα θέματα της ενέργειας. Όπως ξέρετε, οι συνθήκες προβλέπουν όταν υπάρχουν δυσκολίες για την ενεργειακή παροχή, τη δυνατότητα για την Κομισιόν να προτείνει λήψη μέτρων για να λυθεί για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κρίση. Εάν ανακύψει μια τέτοια κατάσταση φέτος το χειμώνα παραδείγματο χάρη, θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα και τι είναι τα, ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα προτείνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα είμαι έτοιμο να δουλέψω μαζί σα για τα TNT, για τα TENI, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργεια και η μεταφορών δεν έχει σημασία. Αν σταθούμε στο θέμα του επερχόμενου χειμώνα. Εγώ πιστεύω ότι ο αντιπρόεδρος κ. Ότιγκερ θα έχει ήδη μια επιτυχία αύριο γιατί μίλησα μαζί του πρώτο έρθω σε αυτή την ακρόαση μου είπε ότι είναι δύσκολε διαπραγματεύσει, αλλά εξακολουθεί να είναι αισιόδοξο ότι μετά από τη σημερινή συνεδρίαση και τη συνέχεια που θα δοθεί αύριο στις Βρυξέλλες θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινό έδαφος, σε ένα κοινό πλαίσιο όπου θα καθοριστούν οι λύσει για αυτό το χειμώνα και το επόμενο έτος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για την Ουκρανία και τη Ρωσία αλλά και για την Ευρώπη. Πιστεύω μια σωστή λύση αυτού του προβλήματος θα καταπραίνει πάρα πολύ τις ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν ιδίω για την αγορά ενέργειας. Τα θετικά νέα τώρα είναι ότι τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής είναι πολύ θετικά και η Ευρώπη γενικά τα καταφέρνει πολύ καλά μπορεί να αντιμετωπίσει έξι μήνες πλήρους αποκοπής από τροφοδοσία από το ρωσικό αέριο, 5-6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για το φυσικό αέριο, που είναι ένα ποσοστό 2-3% της κατανάλωσής μας στο φυσικό αέριο. Βέβαια για ορισμενα κάτι κράτη-μέλη μπορεί να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί εξαρτώνται από το φυσικό αέριο της Ρωσίας πολύ περισσότερο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και αν βρεθούμε σε μια τέτοια έκτατη κατάσταση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στα θέση της και όλες τις εξουσίες της, ώστε να μην επαναληφθούν αυτά που έγιναν το 2009 και δεν θα αντιμετωπίσουμε πάλι μια κατάσταση όπου οι πολίτες στα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα είναι στο σκοτάδι λόγω έλλειψης ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μια κέρια χρονική περίοδο που θα διαμορφώσει και το μέλλον της. και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους στόχους του 2030. Τα ερωτήματα μου είναι πρώτον τι συμπεραίνεται από τα τεστ αντοχής των πυρηνικών σταθμών και πώς η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα και δεύτερον ποια είναι η δική σας προσωπική αντιμετώπιση για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη ως ένα μεταβατικό στάδιο παραγωγής ενέργειας στο δρόμο για μια οικονομία χαμηλή χαμηλής χρήσης άνθρακος. Και δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματιστεί στην Ευρώπη, ευρωπαϊκή πολιτική, από τη γερμανική ενεργειακή πολιτική που είναι κέρια για τις χώρες κεντροανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι τα τεστ αντοχής <clears throat> των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά υπό την έποψη της ασφάλειας και για να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών που στο έδαφος τους υπάρχουν αυτοί οι ποινικοί σταθμοί ότι ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα λοιπόν αυτά τα τεστ αντοχής, ιδίως διότι μπόρεσε έτσι να μεταλαμπαδευτούν βέλτιστες πρακτικές ούτε, ώστε οι πιο σύγχρονες, οι πιο τελευταίες εν πάση περιπτώσει, γνώσεις και εμπειρίες που έχουμε για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες χώρες. Σε 16 χώρες υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί, 14 από αυτές τις χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί οι οποίοι σέβονται τις προδιαγραφές ασφαλείας να μπορέσουν να διατηρηθούν. Στη συνέχεια έχουμε αντιμετωπίσει μια σειρά από σενάρια ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος μέχρι το 2050 και να έχουμε μια μείωση 80 έως 90% μέχρι το ορόσημο του 2050. Τρία από αυτά τα πέντε σενάρια που έχουν αντιμετωπιστεί και μας οδηγούν σε αυτό το στόχο συμπεριλαμβάνουν και την πυρηνική ενέργεια ως πηγή φτωχή σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και αυτή τη στιγμή φυσικά είναι η δεύτερη σημαντικότερη πηγή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να τη θεωρήσουμε ως ένα στοιχείο του ενεργειακού μείγματος που θα συνεχιστεί να είναι σημαντικό στο μέλλον, βέβαια εφόσον ανταποκρίνεται στις ε, ασφαλεία. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεύκοβιτς, όταν μιλάτε για ενεργειακή αποδοτικότητα εννοείται ενεργειακή εξοικονόμηση. Τι θα κάνετε με εκείνες τις χώρες ε, μέλη που θα μπορούσαν ε, να έχουν κάποια προοπτική ανάπτυξη. Δεύτερον, είπατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας ανήκουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν πάνω από 30% μερίδιο. Ε, ε, θα πρέπει και αυτές να υπογραφούν σε εξοικονόμηση ή θα τις εξαιρέσετε. Τρίτον, ε, είπατε ότι ίσως τους ε, ενδεικτικούς στόχους δεν θα πρέπει να τους πάρουμε τόσο σοβαρά. Σημαντικός είναι ο νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου. θέλετε να έχετε μία δεσμευτική οδηγία για το Αιγαίο, για παράδειγμα, για τα ντους ε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει αυτό στην Σκανδιναβία και στην Αυστρία που θα πρέπει να έχουμε νέα τηλέφωνα του ντους, νέες κεφαλές, εκεί όπου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το νερό. Τι θα γίνει με την εφαρμογή μέτρων σε χώρες ε, για τις οποίες δεν έχουν τα μέτρα αυτά απολύτως κανένα νόημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, για το δίλημα που εκφράσατε μεταξύ ενεργειακής ε, αποδοτικότητας και βεβαίως της ε, πίεσης για ενεργειακά αποδοτικούς στόχους. Αλλά όταν το ζητούμενο είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των πολιτικών κλπ, τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά. Βεβαίως μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, αλλά δεύτερο σημαντικό κομμάτι για την αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ε, το eco-design και αν δούμε ε, ποια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα αλλά δεν τα αναφέρουμε συχνά ε, μέχρι το 2020 θα εξοικονομήσουμε το ίδιο ποσό ενέργειας που καταναλώνεται στην Ιταλία σε ένα έτος μόνο με την εφαρμογή της ε, οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού. Και αυτό βεβαίως είναι ένα από τα μέτρα που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και έχουν γελιοποιηθεί από τον τύπο. Αλλά θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα από εδώ. Ε, Υπάρχουν κάποιες τεχνικές ε, μελέτες για τα σεσουάρ ε, μαλλιών και για τις ε, μηχανές ε, καφέ. Ε, και βεβαίως εδώ θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες γιατί αυτό η εξοικονόμηση ενέργεια δεν είναι τόσο σημαντική ώστε να πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς κανόνες. Αλλά όταν μιλάμε για θερμοσύφωνες εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον οικολογικό σχεδιασμό, ούτω ώστε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Ε, και εφόσον το πετύχουμε θα έρθω εδώ ε, και θα σας ε, ρωτήσω, θα ζητήσω και τις προτάσεις για το ποια είναι η καλύτερη προβολή αυτής της πολιτικής και επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μίρια Μντάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή πολιτική η οποία να διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, θα διασφαλίζει την συνέχιση των ενεργειακών πόρων ε, και θα άρει τα εμπόδια αυτών των ε, πασίγνωστων νησίδων ενέργειας που έχουν πρόβλημα διασύνδεσης. Ε, κατά την άποψή σας πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις ε, στις διασυνδέσεις, στις γραμμές παραγωγής, στους θερματικούς σταθμούς. Ποιο είναι το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα στρέφεται προς την ε, Ένωση Ενέργειας και τι θα κάνετε όσον αφορά ε, τις διασυνδέσεις ε, γιατί θα πρέπει όλοι, όλα τα κράτη-μέλη να είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ενέργειας. Είστε από τη Μάλτα νομίζω. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα ε, είναι γεγονός ότι ασχοληθήκαμε πιο πολύ με τις χώρες της Βαλτικής, τη Φιλανδία, με αυτές τις νησίδες ε, ενέργειας. Αλλά έχουμε τέτοιες νησίδες ε, και το είπα και προηγουμένως και στο, στη Νότια Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό γιατί είναι πρόβλημα αλλά είναι ταυτόχρονα και ευκαιρία. αν δει κανεί ε, πώς θα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι πηγές ενέργειας, αν δει κανεί τις ευκαιρίες οι οποίες ε, ε, υπάρχουν όσον αφορά τη δημιουργία ενό μεσογειακού κόμβου ενέργειας, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πραγματικό trading place για το φυσικό αέριο η περιοχή αυτή. Ε, μιλήσαμε προηγουμένως ε, και για τα νέα ε, κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αναφερθήκαμε και στο οικόπεδο Αφροδίτη της Κύπρου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την διαφοροποίηση, τη στρατηγική διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Όσον αφορά τη χώρα σας γνωρίζω την ιδιαιτερότητα της και ένα πρόγραμμα προτεραιότητας ε, ε, στα θέματα και στα προγράμματα κοινών ε, και στο, στον κατάλογο των κοινών προτεραιοτήτων είναι ακριβώς ένα σχέδιο διασύνδεσης της Μάλτας έτσι ώστε η Μάλτα και η Σικελία να, ξεπεράσει, να ξεπεράσουν το, την ενεργειακή τους απομόνωση να ε, βοηθηθεί και η Μάλτα στη διασύνδεσή της με αυτόν τον ενεργειακό κόμβο. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Γκαρντίνη. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Γκαρντίνη. Λοιπόν, πολλά ακούσαμε όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική και οπωσδήποτε ε, ο προβληματισμός μας γενικά αυτή την περίοδο είναι μεγάλος. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη διάσκεψη του Παρισιού το 2015. Ε, μετά την Κοπεχάγη εγώ παρακολουθώ όλες αυτές τις διασκέψεις και πρέπει να πω ότι οι προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί κάθε φορά είναι πολλές και τελικά μετά ε, βλέπουμε ότι έχουν γίνει λίγα. Ε, εγώ άρχισα να ξανά να σκέφτομαι ότι αυτή τη φορά θα είναι η καλή φορά, αλλά παρόλα αυτά ακούω διάφορα πράγματα εντωμεταξύ τα οποία ε, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως δεν θα καταφέρουμε ούτε αυτή τη φορά να υπογράψουμε μια διεθνή συμφωνία η οποία να είναι, συμ, ε, να είναι δεσμευτική. Εδώ μας λέτε διάφορα καινοτομία, ανανεώσιμες αυτές. Τι θα γίνει όμως όσον αφορά τη συλλογική, την συνολική ε, συμφωνία. Αυτά. Και εγώ ε, μοιράζομαι μαζί σας την ίδια αγωνία. Καταλαβαίνω την ε, αγωνία όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και αυτό που λέτε ότι κάθε φορά ξεκινούμε με ε, ε, πολλές προσδοκίες. Ε, είδαμε το πρωτόκολλο του Κιώτο, είδαμε τη διάσκεψη της Βαρσοβίας. Έχουμε πολλές προσδοκίες οι οποίες ενθαρρύνονται από την σκέψη ότι μετά από όσα έχουμε δει να συμβαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη, ότι επιτέλους ε, οι κυβερνώντες ε, θα θα πάρουν αποφάσεις. Ε, ε, αυτή τη στιγμή η αύξηση της ε, θερμοκρασίας είναι 0,8. Αν φτάσει αυτή η αύξηση στους δύο βαθμούς τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Αλλά ταυτοχρόνως βλέπουμε και άλλα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται. Ποτέ δεν είχαμε δει τόσες πολλές φυσικές καταστροφές, ποτέ δεν είχαμε δει τόσο μεγάλες αλλαγές σε πολλές χώρες, γιατί έχουν αλλάξει ε, λόγω της γενικότερης ε, αλλαγής, ε, κλιματικής αλλαγής, πολλά πράγματα και στην Ασία και στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε πλέον αυτή την κριτική μάζα στοιχείων και τεκμηριώσεων, ότι δηλαδή η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικά στοιχεία, ότι μπορεί να έχει πολύ υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος και έχουμε όμως και τα μέτρα και τις δυνατότητες, τις τεχνικές έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, την κλιματική αλλαγή. Πιστεύω λοιπόν ο, επίσης ότι ε, βλέπουμε και κάποιες ε, θετικές εξελίξεις σε χώρες όπως οι Ηνωμένες και η Βραζιλία. Γι' αυτό πιστεύω ότι εάν ακολουθήσουμε μια σωστή τακτική αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα φιλόδοξο συνολικό δεσμευτικό ε, πρόγραμμα. Ο κύριος Κόφορντ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι. Κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, νομίζω ότι μας έχετε δώσει πολύ καλές απαντήσεις απόψε για το πώς να προχωρήσουμε σε μια πράσινη ενεργειακή ένωση στην Ευρώπη αλλά είπατε ότι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι σε επίπεδο ανανεώσιμων ενεργειών στον κόσμο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τις παγκόσμιες επενδύσεις για την καθαρή ενέργεια έχουν μειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες έχουν μειωθεί σημαντικά αυτές οι επενδύσεις. Πρέπει να ξέρω λοιπόν τι <clears throat> πιστεύετε και πώς θα δράσετε συγκεκριμένα ώστε η Ευρώπη να γίνει το νούμερο ένα σε παγκόσμιο επίπεδο για ανανεώσιμες ενέργειες. Τι σημαίνει αυτό, ποιοι είναι οι δομικοί λύθοι αυτής της πρωτοπορίας, πώς μπορούμε να συγκριθούμε με τον υπόλοιπο κόσμο, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ποιο είναι ο στόχος μέχρι το 2030 όταν τον συγκρίνεται με την πραγματικότητα. 27% για ανανεώσιμες ενέργειες είναι φιλόδοξο στόχος για εσάς. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας θέση. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο για τις ανανεώσιμες ενέργειες, γιατί αν δείτε το γεγονός ότι 41% των νέων εγκαταστάσεων για ανανεώσιμη ενέργεια στον κόσμο λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε την ποιότητα της τεχνολογίας μας. Κανείς δεν διαφυσβητεί ότι είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Και αν δούμε τώρα και την επιχειρηματική πλευρά της ποιότητας αυτής, της τεχνολογίας μας, της πράσινες τεχνολογίες. Όλα αυτά καταδεικνύονται από τον ε, από την απασχόληση που δίνει ο τομέα αυτό, την ικανότητα να εξάγουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, το ότι είμαστε ανταγωνιστικοί και μπορούμε να εξάγουμε αυτέ τι πράσινες τεχνολογίες. Πιστεύω λοιπόν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα δούμε να φτάνουμε σε μία, αν θέλετε, κρίσιμη μετάβαση. Θα πετύχουμε την κρίσιμη αυτή μάζα και θα μπορέσει να μειωθεί το κόστος παραγωγή για τι ανανεώσιμε ενέργειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μείωθει λοιπόν σημαντικά. Αν συνεχίσουμε λοιπόν και βελτιώσουμε ακόμα περισσότερε τεχνολογίε, αν δούμε πώ μπορούμε να συνδέουμε τι ανανεώσιμε ενέργειε στο δίκτυό μα και αν ξεπεράσουμε τα σημεία συμφόρηση, μπορούμε έτσι να υποφελθούμε πολύ περισσότερο από την ενέργεια, τι ανανεώσιμε ενέργειε, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνέ επίπεδο και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα που εξηγεί γιατί πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για την ανανεώσιμη ενέργεια και αυτό θα οδηγήσει στην επίτευξη ενό στόχου 27% και περισσότερο από 27% γιατί η εμπειρία μα με τι επιχειρήσει και την τεχνολογία θα μας οδηγήσουν σε πολύ περισσότερη χρήση ανανεώσιμων από 27% κύριος Βέρνετ Λάγκελ. Κύριε Σέρκοβιτς. Δεν απαντήσατε ουσιαστικά το ερώτημα της κυρίας Κιώστιγκερ για το ποια θέση πήρατε όταν αποφάσισε ο κύριος, όταν πρώτο ο κύριος Αλμούνια να πάρουμε, πάρει η Επιτροπή μια θέση για τον Λοιπόν, Ψήφισατε υπέρ ή κατά. Δεν πρόκειται για τη θέση σας για την πυρηνική ενέργεια. Μιλάμε για μια τεράστια στρέβλωση ανταγωνισμού. Πάνω από 35 δισεκατομμύρια χάνονται για την Ευρώπη γιατί υπάρχουν εγγυήσεις για τιμή πυρηνικής ενέργειας πολύ πάνω από τις τιμές αγοράς. Μιλάει τώρα η Κομισιόν για βιοκαύσιμα προ γενιάς που θα υποστηρίζεται μέχρι το 2020. Έχετε και την οικολογική σχεδίαση. Αλλά τι κάνετε με την Γαλλία, τι κάνετε με τη Γαλλία, μαζί ζητήσει τα ίδια πράγματα όπως η Μεγάλη Βρετανία για την πυρηνική ενέργεια. Ουσιαστικά λοιπόν φεύγει από το παράθυρο όλη η στρατηγική σα για την ανανεώσιμη ενέργεια, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη όταν ήδη σε μια τέτοια περίπτωση όπως τη Μεγάλη Βρετανία έγινε ένα τόσο μεγάλο σφάλμα. Αυτό έγινε μετά από την εκλογή του Γιούκερ και όχι πριν κιόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στεναρή αυτή δήλωση που κάνετε. Αν ξανάφουμε και πάλι σε μια περίπτωση όπως το, η περίπτωση του Χίνκλεϊ. Σας λέω ότι αυτό δεν ήταν ένα θέμα που αντιμετωπίστηκε ως θέμα ενεργειακών επιλογών. Ήταν ένα θέμα ανταγωνισμού και αντιμετωπίστηκε από τους κέριους οικονομολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και ήταν σαφές εδώ ότι μιλούσαμε για τον κίνδυνο μιας αστοχία στην αγορά και ότι ήταν απαραίτητη η κρατική βοήθεια για να διατηρηθεί. Ναι, και αν με ρωτάτε, εγώ ψήφισα υπέρ αυτού του μέτρου, γιατί θεώρησα ότι ήταν πλήρε συμβατό με του κανόνε ανταγωνισμού για τι κρατικέ επιδοτήσει και σε αυτή την περίπτωση εάν δεν σεβόμασταν τους κανόνες ανταγωνισμού που προέρχονται από τις συνθήκες, η Κομισιόν δεν θα δεχόταν, δεν θα εφάρμοσε σωστά τη συνθήκη και όλα αυτά που προδιαγράφει για τις κρατικές επιδοτήσεις. Για τα βιοκαύσιμα, ο λόγος για τον οποίο εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τους στόχους για τα βιοκαύσιμα ως το 2020 είναι γιατί απογοητευτήκαμε από την πρώτη γενιά βιοκαυσίμων που είχαν ε, συνέπειες απρόβλεπτες. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ε, ουσιαστικά εκτόπισαν την παραγωγή τροφίμων για να γίνει παραγωγή βιοκαυσίμων. και τα καύσιμα αυτά και η παραγωγή του τη πρώτη γενιά δεν είχαν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε σε επίπεδο μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. Επομένω, οι προτάσει μα για την έμεση αλλαγή χρήση γη, στο iLook, και να μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτό το θέμα ε, είναι προτάσει που θα πρέπει να υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων. Ναι, ε, κύριε Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο από το παλαιό σύστημα ενέργειας με τα μεγάλα ε, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, ε, πυρηνικής ενέργειας, τα, στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Ε, βεβαίως εδώ υπάρχουν πολλές τριβές σε ορισμένε χώρες. αυτοί που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα επιθυμούν επιδοτήσεις για τη λειτουργία των εργοστασίων τους πώς ε, θα, πώς μπορείτε να εμποδίσετε ότι υπάρχουν 28 τέτοια εργοστάσια που ζητούν επιδοτήσεις. Δεύτερον, όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, χαίρομαι που υπερασπιστήκατε την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, γιατί εδώ υπάρχει ευρύ πεδίο για ε, λαϊκισμό και δημαγωγία. Ε, ε, η πρόταση, η Επιτροπή έχει προτείνει και 17 άλλα προϊόντα για να συμπεριληφθούν ε, στην ε, ρύθμιση του, του eco-design. Σας συμφωνείτε με αυτές τις προτάσεις. Απάντηση. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση και στρεφόμαστε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν χώρες ε, που έχουν ε, πολύ ηλιοφάνεια και αιωλική ενέργεια. Ε, από την άλλη η συσσόρευση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί, η συμφόρηση της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, προβλήματα στο δίκτυο δηλαδή. Ε, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση των συστημάτων ε, μετάδοσης ε, ενέργειας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Γιατί, και πιστεύω ότι αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο κλειδί για μια καλύτερη ολοκλήρωση και συμπερίληψη ανώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημά μας. Ε, ε, ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξορρόπηση στα δίκτυα. Όσον αφορά το eco-design και τη σχετική οδηγία, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε, αλλά με έναν έξυπνο τρόπο, δηλαδή να βασίσουμε τις προτάσεις μας σε πολύ στέρεες επιστημονικές αναλύσεις και να εμπιστευτούμε μόνο εκείνους τους τομείς όπου είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, θα υπάρχει προσθέμενη αξία και θα αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Ε, και ε, επίσης το εξή. Αυτό που χρειαζόμαστε εδώ είναι πιο έντονες ε, διαβουλεύσεις με τους πολίτες ακριβώς λόγω του όγκου γραφειοκρατίας ε, και λόγω του στόχου ε, εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους για τους πολίτες. Ο κύριος Νούνο Μέλου, τελευταία ερώτηση. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, υπάρχουν πολλές απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, τρομοκρατικές επιθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί ότι πρέπει να καλύπτει μονάχα λιγότερο από το 50%. Ένα μεγάλο μέρος από τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καλύπτονται από εισαγωγές και φτάνει η συνολική, το συνολικό κόστος σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί λοιπόν, σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ μάλλον, ποιοι είναι οι μηχανισμοί ασφάλειας που προβλέπετε για τη ε, διαμετακόμιση φυσικού αέριου. Όταν ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Ιβυρική Χερσόνησο, θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένες οι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ή όχι. Thank uh, ευχαριστώ. Ε, η ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, ε, είδαμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής ότι είμαστε σε καλύτερη θέση, σε πιο ισχυρή θέση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Ωστόσο, ε, και πρέπει και, μπορούμε αλλά και πρέπει να ε, βελτιώσουμε την ε, κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως και ποια είναι τα εθνικά προγράμματα, ποια είναι, αν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων. Επίσης να δούμε τι δυνατότητες αποθήκευσης έχουμε γιατί και εδώ μπορεί να υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και εν πάση περιπτώσει τα ε, κυρίαρχα ε, ζητήματα και τα κυρίαρχα στοιχεία όσον αφορά τις διαμεθοριακές συνδέσεις, όσον αφορά τις ανάδρομες ροές. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη έτσι ώστε να βρούμε και να δημιουργήσουμε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο που θα είναι σε θέση να βοηθήσει όποια χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα επίγοντα τα ε, σχέδια τα οποία, στα οποία αναφέρεστε είναι σχέδια τα οποία έχουν ε, ήδη καταρτιστεί και από τις ε, χώρες μέλη. Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος για τις περιοχές αυτές οι οποίες οι οποίες πιέζονται περισσότερο ε, νομίζω ότι αρχικά η διευκόλυνση Connecting Europe όντως ήταν πολύ πιο ε, φιλόδοξη και είχε και μεγαλύτερη προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες ε, και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και την βοήθεια των ιδιωτικών φορέων έτσι ώστε και στην, στις διασυνδέσεις του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου να έχουμε ε, τα καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Μετά από την τελευταία απάντηση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή συζήτηση για τις ερωτήσεις τους. Να ευχαριστήσω βεβαίως ε, και τον υποψήφιο επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να ε, δώσω το λόγο στον υποψήφιο ε, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να κάνει την τελική του τοποθέτηση η οποία δεν θα πρέπει να υπερβεί τα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι η ώρα περνάει και πρέπει να τελειώσετε. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας, γιατί νομίζω ότι επιβεβαίωσαν την πραγματογνωμοσύνη σας. Ε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Έρευνας. Επομένως, διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά και και τις γνώσεις σας αλλά και την αφοσίωση που έχετε όσον αφορά ε, τα ζητήματα αυτά που μας ε, απασχολούν. Ξέρω ότι εργάζεστε ε, πολλά χρόνια εδώ και πολλά χρόνια ε, για τα θέματα αυτά και ε, έχετε πραγματικά επιτύχει πάρα πολλά. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η επιτυχία και η σε αντιμετώπιση των ζητημάτων συνεχιστεί και τα επόμενα πέντε χρόνια στη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Προσπάθησα να σας εξηγήσω ποια είναι τα κριτήρια ε, ε, με τα οποία κρίνουν και εμάς και την Επιτροπή δηλαδή και τους, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πολίτες και επ' να βασίσω και τους πυλώνες εργασίας μου Θέλουν οι πολίτες λοιπόν καθαρή ε, προσιτή ενέργεια. Αυτό πρέπει να τους δώσουμε. Επίσης ζητούν αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη και ε, ασφάλεια όσον αφορά την ε, ενέργεια. Όσον αφορά τώρα την ανάπτυξη θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αντιμετωπίζει η Ευρώπη πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, σκληρό άγριο ανταγωνισμό σε αυτόν τον νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Θα πρέπει να το κάνουμε ε, με τρόπο σωστό, ε, έτσι όπως εμείς καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη, δηλαδή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον ε, και με διατήρηση των κοινωνικών προτύπων. Φυσικά δεν υπάρχουν εύκολες ερωτήσεις σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα και ε, νομίζω ότι ο τρόπος που θα μας αντιμετωπίσουν οι πολίτες, ε, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι κριτές, ε, θα είναι και ο, τρόπο, θα είναι και ο οδηγός μας σε αυτήν την, σε αυτή την πορεία. Πιστεύω πάντως ότι η Ευρώπη είναι στη, σε σωστή θέση, έχει όλα αυτά τα απαραίτητα συστατικά έτσι ώστε να προχωρήσει και πιστεύω ότι εάν καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού θα καταφέρουμε να καλύψουμε τις διαφορές. Ξέρετε ότι στην παρούσα θητεία της Κομισιόν ήμουν υπεύθυνο και για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο ε, και δούλεψα πάρα πολύ, συνεργάστηκα πολύ με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, την Νομική Επιτροπή, πολύ στενά συνεργάστηκα με τον ε, Πρόεδρο Μπούζεξ, τη διάσκεψη των ε, Προέδρων. και την εποχή βεβαίως που ήταν και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, εγώ είμαι θερμός υποστηρικτής της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων, είμαι θερμός υποστηρικτής του δομημένου διαλόγου, αλλά και της ε, σωστής ε, αξιολόγησης, προετοιμασίας ε, της εργασίας. Και όσον αφορά και εάν εγκρίνεται την νέα μου θέση, θα συνεχίσω την συνεργασία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα είμαι πάντα έτοιμος να έρθω εδώ οποτεδήποτε μου το ζητήσετε να συζητήσω μαζί σας, να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και βεβαίως και σε επίσημο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο με τον καθένα από εσά θα ήθελα να έχω ε, την ε, επαφή αυτή η οποία θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και εάν ε, τύχω τη στήριξή σας ε, δεσμεύομαι να συνεχίσω την καλή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε και για τις δηλώσεις σας ε, και για τις απαντήσεις και για αυτές τις πέντε μέρες σκληρής δουλειάς που κάνατε έτσι ώστε να προετοιμαστείτε για την ακρόαση αυτή. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι εδώ σας ευχαριστούν. Σας ευχαριστώ και εγώ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί έχετε υπομονή αλλά έχετε και πάθος. Είσαστε παθιασμένοι με τα θέματα. Και σε ό,τι αφορά την Ήτρε, οι συντονιστές για την συνάντηση αξιολόγησης θα συναντηθούν αύριο στις 9.30. Με, μετά θα γίνει κοινή μας συνεδρίαση με την Επιτροπή Ήτρε ε, Ευχαριστώ πολύ και τον Τζάνι Λαβία. Και εγώ ευχαριστώ. Αύριο θα έχουμε τη συνάντησή μας στις 9 και μετά θα συναντήσουμε και τους συντονιστές της Επιτροπής Ήτρε για την τελική μας αξιολόγηση. Ε, καλή όρεξη λίγο αργά είναι, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Γεια σας.